Κυρίε και κύριοι, ίσω μπορούμε να αρχίσουμε. Θα ήθελα να σα χαιρετήσω όλου στην καρδιότητα. Να περάσω στο σημείο ένα ημερησίας διάταξη, δηλαδή την ε, έγκριση τη σημερινή διάταξη αυτή. Έχετε την ημερησία διάταξη μπροστά σα, το προσέδιο ο πρόεδρος του Προέδρου της Επιτροπής Επιστήμης και Τεχνολογίας τον ΗΠΑ μεριώθηκε γιατί δεν μπορεί να είναι παρόν. Και γράφουμε από αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης, δηλαδή οι συντονιστές αρχίζουν στην εδρίασή τους αμέσως μετά το τέλος της ακρόασης. Αν δεν υπάρχουν άλλες επιθυμίες ε, ε, για την ημερησία διάταξη την εγκρίνουμε. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Άλλος κανένας δεν έχει κάτι να πει, δεν έχω καμία πληροφόρηση να σας δώσω. Έχετε τα πρακτικά της συνεδρίας μπροστά σας, των συνεδριάσεων μάλλον. Εάν δεν έχετε καμία παρατήρηση μπορεί να εγκριθούν. Περνάμε στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης, μήνυα ακρόαση για την ασφάλεια φοδιασμού με αέριο φυσικό. Πριν από αρκετό καιρό είχαμε αποφασίσει να οργανώσουμε μια ακρόαση για το θέμα για να το εξάσουμε λεπτομερέστερα. Έχουμε την έρευνα και πρόταση κομισιών που θα θέλουμε να σκεφτούμε καλύτερα μέσα στις πλαίσια μιας βιομηχανικής πολιτικής. Έχουμε καλέσει διάφορους εμπειρογνώμονες. Έχουμε λοιπόν και τον ειδικά υπεύθυνο αντιπρόεδρο και εισηγητή του Κοινοβουλίου, τον κύριο Βίταλ Κβάντας. Θα ήθελα να χαιρετήσω του εμπειρογνώμονε, τον κύριο Μπόρτς, ο οποίο δυστυχώ δεν μπόρεσε να έρθει. Ήρθε ο κύριο Στέρτσερ, ανταυτού, ο κύριο Άντφαν Μπούμετα, ο κύριο Μάρσελ Κράμα και ο καθηγητή Όλιβερ Μπέτσουγε. είχαμε συμφωνήσει κάθε προγνώμενος να έχει περίπου 15 λεπτά στη διάθεσή του για να κάνει μια παρουσίαση και μετά μπορέσουμε να περάσουμε στην ακρόαση. Εκτός αν ο κύριος Βιταλκβάτρας, εισαγωγικά θα ήθελε να κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Όχι, ωραία. Μπορούμε λοιπόν να αρχίσουμε με τη σειρά που έχετε μπροστά σας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μιχαήλ Σμέλτσερ πρώτο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή. Είμαι σήμερα εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ρυθμιστικών Αρχών ε, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Εγώ δουλεύω για την e-control, την ε, Αυστριακή Ρυθμιστική Αρχή το διευκρινίζω γιατί έχει διαφορετικό ρόλο από τις άλλες ρυθμιστικές αρχές. Στην Αυστρία είναι υπεύθυνη η αρχή και για κάποιες πτυχές της ασφάλειας εφοδιασμού για την πρόληψη κρίσεων, οπότε πρέπει να έχει ένα σχέδιο πρόληψης κρίσεων και είναι υπεύθυνο και για την επιτήρηση. Και με βάση αυτή την εμπειρία είναι και η παρουσίασή μου. Εάν ε, δείτε την κατάσταση που είχαμε στην αρχή του έτους, τις πρώτες δύο εβδομάδες του Ιανουαρίου και τα μαθήματα που αντλήσαμε, Βλέπουμε πως είναι σημαντικό να έχουμε μια εσωτερική αγορά αερίου που θα λειτουργεί. Επίσης κάποιες χώρες στην Ευρώπη, ειδικά στην Νοτιοανατολική Ευρώπη που δεν είναι διασυνδεδεμένες, ε, τα προβλήματα ήταν μεγαλύτερα από ότι σε άλλες χώρες όπου οι αγορές είναι διασυνδεδεμένες και άρα ήταν πιο εύκολο να υπάρξει ένα σύστημα πιο ευέλικτο μεταφοράς αερίου. Επίσης, στην κατάσταση αυτή που είχαμε στην αρχή του έτους είδαμε πως είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να αγοράζουν σε υγροποιημένη μορφή το αέριο οι πελάτες από άλλους προμηθευτές οπότε είναι η σημαντικότερη εγγύηση απρόσκοπτης ροής η λειτουργούσα εσωτερική αγορά επίσης με βάση την αυστριακή εμπειρία είδαμε πως είναι καλύτερο να αφήσουμε την αγορά να λειτουργήσει όσο το δυνατόν περισσότερο γιατί στην κατάσταση αυτή οι προμηθευτές και οι διαχειριστές του δικτύου βρίσκουν πολλές λύσεις για να αντιστρέψουν τις ροές και ε, δεν χρειάζεται να αρχίσουμε αμέσως με κρατικές παρεμβάσεις γιατί τότε βεβαίως σταματά κάθε λειτουργία από αυτού που συμμετέχουν στην αγορά. Σημαντικό λοιπόν είναι να αφήσουμε την αγορά να λειτουργήσει όσο είναι δυνατόν, αλλά να υπάρχει και μια γενική εικόνα για την ασφάλεια προμήθεια, να υπάρχει δηλαδή μια εικόνα για το ποια είναι η ζήτηση και η προσφορά. Σε μια τέτοια κατάσταση όπως αυτή που είχαμε την αρχή του έτους είναι πάρα πολύ χρήσιμη μια γρήγορη ευρωπαϊκή απάντηση όταν έχουμε κρίση. Σημαντικό είναι να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση στις διάφορες ε, χώρες, να υπάρχει μια γενική εικόνα όπως σας είπα και οι χώρες να βοηθάνε η μία την άλλη. Οπότε ως ε, Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Εθνιστικών Αρχών καλωσορίζουμε την πρόταση της Κομισιόν για έναν ε, σχετικό κανονισμό. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που είναι ουσιαστικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε σαφή ορισμό των ρόλων και των ευθυνών των αρμοδίων αρχών ε, όχι μόνο αυτών βεβαίως αλλά και όλων ε, όσων συμμετέχουν στην αγορά είναι σημαντικό να έχουμε προληπτικό σχέδιο δράσης ε, να ξέρουμε λοιπόν ποιος είναι ο ρόλος και ευθύνη του καθενός ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι να υπάρχει ένα πρότυπο υποδομών και προμήθειας όπως είδαμε στην αρχή του έτους, δεν είχαμε πανευρωπαϊκή κρίση γιατί υπήρχε πολύ αέριο στη Βόρεια Ευρώπη αλλά το ζήτημα ήταν πώς θα φτάσει το αέριο στις χώρες εκείνες που είχαν το πρόβλημα. Οπότε ένα πρότυπο, μια προδιαγραφή για την υποδομή είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ της ε, προδιαγραφής ε, υποδομών και προμήθειας και για να έχουν και όλοι οι την ίδια κατάσταση όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν σαφή βήματα για να πάμε προς την κατεύθυνση της ε, κινητικοποίησης και όπως σας είπα πρέπει να αφήσουμε την αγορά να λειτουργήσει όσο μπορεί και μόνο εάν δεν μπορέσει η αγορά να δώσει λύση τότε ε, είναι απαραίτητη η παρέμβαση των κρατών. Επίσης σημαντικό είναι να υπάρχει ένα σχέδιο προληπτικό και σχέδιο εκτάκτου ανάγκης, κάτι το οποίο έχουμε προετοιμάσει στην Αυστρία από το 2006, όταν είχαμε συζητήσει με όλους τους φορείς της αγοράς αυτό το προληπτικό σχέδιο δράσης και ήμασταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που είχαμε τέτοιο σχέδιο γιατί κάθε ρόλος και ευθύνη είχε καθοριστεί στο σχέδιο εκτάκτου ανάγκης και νομίζω πως η πρόταση να υπάρξει ένα συντονισμό σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο είναι πολύ σημαντική. Επίσης, ο ρόλος της ομάδας συντονισμού αερίου είναι πολύ σημαντικός γιατί εκεί μπορεί να συντονιστούν τα μέτρα, να ανταλλαχθούν τα δεδομένα για να ενισχυθεί ο ρόλος ε, των αρχών συντονισμού. Εκεί που θεωρούμε ότι χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις είναι στο ότι θεωρούμε πως μπορούν να εμπλακούν στην κατάρτιση προληπτικών σχεδίων και σχεδίων εκτάκτου ανάγκης οι ρυθμιστικές αρχές. Εμείς είχαμε εμπειρία σχετική στην Αυστρία γιατί είναι οι ρυθμιστικές αρχές ε, πολύ κοντά στην ε, αγορά οπότε η ανάμειξή τους ε, είναι πολύ σημαντική. Επίσης, θεωρούμε πως ε, θα πρέπει να υπάρξει μια κοινοποίηση για την υποχρέωση αντιστροφής της ροής. Ε, μπορούν να γίνουν κάποιες εξαιρέσεις για τους αγωγούς εκείνους που είναι συνδεδεμένοι με τον παραγωγό, με την παραγωγή και άρα εκεί όπου δεν γίνεται να αντιστραφεί η ροή πρέπει να το διευκρινίσουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικές οι υποχρεώσεις ε, αντιστροφής της ροής, ειδικά με αυτά τα οποία είδαμε στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Θεωρούμε επίσης πως πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω το κόστος, γιατί μιλάμε για επενδύσεις στις υποδομές, από τις οποίες επενδύσεις επωφελείται ένα άλλο κράτος Οπότε σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσει ποιος είναι υπεύθυνος για αυτές τις επενδύσεις και πώς θα είναι η κατανομή του κόστους. Ένα άλλο ζήτημα που είδαμε στην αρχή του έτους είναι η παραγωγή του ηλεκτρισμού και η και η περιφερειακή θέρμανση Ίσως ε, οι προστατευόμενοι πελάτες να περιοριστούν π.χ. στα νοικοκυριά, αλλά και η παραγωγή του ηλεκτρισμού και οι ανάγκε θέρμανση είναι πάρα πολύ σημαντικά κριτήρια για τη διαχείριση κρίσεων. Επίσης θεωρούμε πως ε, θα πρέπει να υπάρξει ένα υψηλότερο κατόφλι για μια κοινοτική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Βλέπουμε πως τα εθνικά και τα περιφερειακά σχέδια εκτάκτου ανάγκης είναι πιο αποτελεσματικά από το να έχουμε ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τώρα επανέρχομαι στις επενδύσεις αντιστροφής της ροής που είναι πολύ σημαντικές για κάποιες ε, περιοχές που επηρεάστηκαν από την κρίση στην Ευρώπη. Αν δούμε τις επενδύσεις αυτές στην νοτιοανατολική Ευρώπη υπολογίζεται πως θα είναι γύρω στα 80-90 εκατομμύρια ευρώ. Εάν δούμε ποια ήταν η οικονομική ζημία στις χώρες αυτές, όπως ε, την ανέφεραν οι αρχές, μιλάμε για 700-800 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε νομίζω είναι σημαντικές αυτές οι επενδύσεις γιατί δεν είναι τόσο υψηλές, αλλά θα αντιμετωπίσουν πολύ καλύτερα μια τέτοια κατάσταση. Τι άλλο χρειάζεται τώρα για τις μελλοντικέ κρίσεις παροχής αερίου. Αυτό το οποίο βλέπουμε και καλύπτεται και από άλλους ε, κανονισμούς. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια. Βλέπουμε για τις ε, χώρες εκείνες που δεν επηρεάστηκαν άμεσα από την κρίση πως είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι τα αποθέματα Οπότε χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια, να ξέρουμε ποιες είναι οι πραγματικές ροές αερίου. Οπότε και εδώ πέρα χρειάζεται διαφάνεια, όχι μόνο για τον ανταγωνισμό, αλλά και για την ασφάλεια εφοδιασμού. Επίσης, καλύτερη πρόσβαση σε ευέλικτο αέριο, στην αγορά δηλαδή να χρησιμοποιηθεί καλύτερα η υποδομή, καλύτερες ε, δυνατότητες και καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Βλέπουμε πως ε, μετά από 10 μέρες έφτασε το αέριο από τη Βόρεια Ευρώπη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αν υπάρχει λοιπόν μια πιο συντονισμένη διαχείριση των υποδομών θα λυθεί πιο εύκολα μια τέτοια κατάσταση. Επίσης πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση των υποδομών, δηλαδή αν υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική ενέργειας, πώς θα είναι αυτή, μπορούμε να στραφούμε σε νέες πηγές, στη Μέση Ανατολή, πώς θα έρθει όμως από εκεί το αέριο στην Ευρώπη. Επίσης, θα μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερο βάρος στην εγχώρια παραγωγή, π.χ. με κάποιες μη συμβατικές πηγές αερίου είχαν κάποια επιτυχία οι Ηνωμένε Πολιτείες και βεβαίως πρέπει να έχουμε και προγραμματισμένες επενδύσεις ε, είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόταση του εκαετούς ε, επενδυτικού προγράμματος, αλλά πρέπει να υλοποιηθούν και όλες αυτές οι επενδύσεις. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για όσα μας είπατε και για το γνώστο ότι ήσασταν πραγματικά σύντομος και ακριβής. Αυτά μας βοήθησαν. Επόμενος έχει ο κύριος Άτφαν Μπαέμ, επικεφαλής της ε, τους ε, ε, Διεθνούς ε, Υπηρεσίες Ενεργείας. Έχετε το λόγο. Okay. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση, πεντάλεπτη ας πούμε, για την Ευρωπαϊκή Αγορά Αέριο και για το συμβάν του περασμένου Ιανουαρίου και μετά θα αφιερώσω 10 λεπτά σε συγκεκριμένα σχόλια για τον εν λόγω κανονισμό. Κάποιε διαφάνειες πρώτα απ' όλα για το που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την παραγωγή φυσικού αερίου στην Ευρώπη σε σχέση με άλλες παραγωγές του κόσμου, περιοχές παραγωγής του κόσμου. Η παραγωγή 2006-2030 θα βλέπει ότι στην Ευρώπη του ΩΣΑ, στην Νορβηγία δηλαδή, από 300 θα πάμε σε 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Αν το συγκρίνετε αυτό με τη ζήτηση του 2030, θα δείτε ότι η ιστορική αγορά α, χωρίς την Νορβηγία 100 θα είναι το 2030, το οποίο σημαίνει ότι αυξάνεται η ζήτηση και άρα η πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη για την κάλυψη της ε, ζήτησης στην Ευρώπη. Τα αριθμητικά αυτά ποσά έχουν επικαιροποιηθεί το καλοκαίρι θα δούμε και αύριο κάποια νέα στοιχεία, ίσως κάπως διαφορετικά από τα σήμερα, αλλά δεν μπορώ να τα αποκαλύψω σήμερα. Θα τα δείτε αύριο στον τύπο. Αυξημένη <clears throat> πάντως είναι η ζήτηση και μειωμένη η παραγωγή. Αυτό είναι το μήνυμα. Τώρα για τις διαταραχές. 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου απολέστησαν στην Ευρώπη και άλλα 2 δις στην Ουκρανία από μόνη της. Το πρόβλημα λύθηκε από την εμπορική αποθήκευση 75% από τις ευρωπαϊκές χώρες, Ιταλία, Αυστρία, Ενωμένο Βασίλειο, κάποιες περαιτέρω τροφοδοσίες από τη Ρωσία, από το LNG και από άλλες ε, χώρες ε, παραγωγής όπως η Νορβηγία και οι χώρες. Όπως είπε και ο προλαλής σας, χρειάστηκε χρόνο στην αγορά για να αντιδράσει την πρώτη μέρα της κρίσης ήδη η αγορά αντέδρασε. Ίσως ό,τι αφορά ιδιαίτερα το σημείο σύνδεσης, διασύνδεσης ε, του Νομεροσυλίου με το Βέλγιο. Και έναν εναλλακτική τρόπη και διαδρόμες η Γερμανία και η Κροατία μετά από μέρες χάρη στην Τουρκία μπόρεσαν να εγκρίνουν κάποιες εναλλακτικέ διαδρομές. Πάντως χρειάστηκε πάνω από μια εβδομάδα ε, για την ε, Σερβία και τη Βοσνία μέσω Ουγγαρία να περάσει η τροφοδοσία και φτάσαμε στο τέλος της κρίσης ουσιαστικά μέχρι να λειτουργήσει το μέτρο της αντίστροφης ροής από την Ελλάδα στη Βουλγαρία για παράδειγμα. Αυτό για να καταδείξουμε τις δυσκολίες που έχουμε με την αντιστροφή ροή, <clears throat> όχι μόνο τις δυσκολίες τεχνικής φύσεως, για την αντιστροφή δηλαδή των αγωγών, αλλά και τις δυσκολίες που υπάρχουν στα συμβόλαια, στις συμβάσεις. Με τις επιχειρήσεις ε, που ε, δρούν στον τομέα δεν έχουν συνηθίσει την αντιστροφή, οπότε θα έπρεπε να συναυθούν νέες συμβάσεις, κατά το οποίο ήταν χρονοβόρο. Ήταν λοιπόν σημαντικό το δίδαγμα και για τον επόμενο χειμώνα, για τον χειμώνα που έρχεται, έχουμε ετοιμαστεί, έχουν γίνει επενδύσεις στις αντίστροφες ροές. Είμαστε πιο έτοιμοι τώρα, έχουμε κάποιες ε, συμβάσεις για αντίστροφες ροές και αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ καλό και χρήσιμο. Τώρα, δύο λόγια για τον κανονισμό αυτό καθεαυτό. Είχαμε μια υπουργική διάσκεψη στον IEA στις 14 και 15 Οκτωβρίου. Οι Υπουργοί μίλησαν για την ασφάλεια στον αγορά αερίου και έκαναν μια σαφή δήλωση με τρία σημεία. Πρώτον, ορθά λειτουργούσα αγορά, που είναι ο καλύτερος τρόπος ε, υπερβασής των προβλημάτων. Δεύτερον, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να επαναξιολογήσει τις πολιτικές του και να βελτιώσει την ετοιμότητά του. Και τρίτον, η ΑΕΕ, η Γραμματεία στο Παρίσι, παρακολουθεί την κατάσταση όλων των κρατών μελών και θα περιλάβει τις διατροχές στο φυσικό αέριο σε ασκήσεις προσωμείωσης και αναθεώρησης ούτως ώστε να συλλέξει τις απόψεις όλων σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος της παράθεσης. Οι υπουργοί μας λοιπόν σημείωσαν ότι το φυσικό αέριο εξελίσσεται από μια τοπική αγορά προς μια σφαιρική παγκόσμια αγορά όπου η LNG θα μπορούσε να είναι διαμεσολαβητής, διαιτητής. Το είδαμε αυτό το τελευταία χρόνια και ως συνέπεια οι τοπικές διαταραχές μεταγγίζονται, επηρεάζουν και άλλες περιοχές. Η ΑΕΕ έχει ένα καλό σύστημα για την καταπολέμηση των διαταραχών αυτών, των βασικών κανονισμών, αλλά και συλλογήσουν συλλογήσεων των χωρών και προσωμιώσεων. Η απόφαση για μια συλλογική δράση για την ΑΕΕ για το πετρέλαιο λήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου όλες οι χώρες αντιπροσωπεύονται και ένα αίτημα μπορεί να υποβάλει ή ο εκτελεστικό διευθυντή το οποιαδήποτε χώρα μέλο του ΑΕΕ επί τη βάση τη αξιολόγηση που έγινε. Έχουμε τακτικέ ασκήσει για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η απόφαση μπορεί να ληφθεί εντό 24 με 48 ωρών. Εφόσον 19 από τα 28 μέλη του ΑΕΕ είναι και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υπουργοί μα, όπω είπα προηγουμένω, σαφώς θέλησαν να αποφύγουν επικαλύψεις ε, της εργασίας του ΑΕΕ με τι ε, τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε δεν υπάρχει ε, περίπτωση να προκύψει κανονισμός της ΑΕΕ για την ασφάλεια στο φυσικό αέριο τα επόμενα, τα μέσα επόμενα τουλάχιστον χρόνια. Θα αναμένουμε τις εξελίξεις. Το σχέδιο κανονισμού που βρίσκεται επιτάπητο σήμερα είναι πολύ λεπτομερές και πυροδοτεί πολλές τεχνικές και πολιτικές συζητήσεις. Θα προσπαθήσω να κάνω κάποια γενικά σχόλια για τέσσερα ζητήματα κλειδιά. Δομές, υποδομές, τροφοδοσία, ε, ηλεκτρική ενέργεια και οργανωτικές ικανότητες για ταχεία αντίδραση σε περίπτωση διαταραχής. Όμως γενικά με τον ΑΕΕ είμαστε θετικοί, είμαστε, ε, σαφώς πιστεύουμε ότι είναι πολύ θετικό αυτό το βήμα που γίνεται μέσω του κανονισμό για τις υποδομές. Για να είμαστε σε θέση να παραδώσουμε φυσικό αέριο στις ποσότητες που ζητούν οι συμμετέχοντες στην αγορά, οι υποδομές θα πρέπει να αντέχουν τις αποτυχίες το, ένα, το ω ένα ως κριτήριο είναι το πιο σωστό, δεν θα μπω σε λεπτομέρειε. αλλά έχω πέντε σχόλια, πέντε λέγω σχόλια επί της προτάσεως κανονισμού για το, 1, μειον, για το N 1. Είναι σαφέ ότι ο κανονισμό το υπολογίζει αυτό επί τη βάση των ανώτατων όγκων. Οι ανώτατοι όγκοι θα πρέπει να είναι αρκετοί. Δεν χρειάζεται να έχουμε αποθέματα εάν αυτή η δυνατότητα η δεν χρησιμοποιείται ποτέ. Δεύτερον, ε, το 1 1 είναι ένα κριτήριο που ισχύει για όλους. Δεν χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει αυτό το περιθώριο, η προθεσμία των 60 ημερών. Τρίτον, τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να αφορούν και τη διέλευση. Οι γείτονες χώρες ε, είναι ελεξαρτούμενες αλλά όχι για τη συνολική δυνατότητα διέλευσης, μόνο για τα συμβόλαια διέλευσης πρέπει να ισχύει κάτι τέτοιο. Και τέταρτο, μέτρα από την πλευρά της ζήτησης μπορούν να τροποποιήσουν ενδεχομένω τον κανόνα 1-1. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό δημιουργεί σύγχυση. Το πρότυπο για τις υποδομές θα πρέπει να αποτελεί διασφάλιση για την παράδοση όλων των ποσοτήτων που προβλέπονται από τα συμβόλαια. Για την αποθήκευση πολύ σημαντική. Όπω είδαμε με την τελευταία κρίση του Ιανουαρίου, 75% τη κρίση. μπορέσαμε, ε, ε, υπερπηδήθηκε λόγω τη αποθήκευση. Ήμασταν τυχεροί λοιπόν, γιατί η ζήτηση ήταν χαμηλή λόγω τη ύφεση και η αποθήκευση ήταν στο απόγειό διότι ήμασταν στην αρχή του χειμώνα. Το πρόσθετο αέριο κυρίω ήρθε από την εμπορική αποθήκευση όπω είπα, αποθήκευση που στόχο έχει την εξάντληση των αποθεμάτων αυτών μέχρι τα τέλη του Ιουνίου. Αν είχαμε λοιπόν την κρίση τα τέλη Μαρτίου τι θα είχε γίνει. Η στρατηγική αποθήκευση και ο έλεγχο των κυβερνήσεων θα μπορούσαν να είναι μια εναλλακτική αποθήκευση ιδιωτική, μάλλον ε, κρατική, κυβερνητική ή θα μπορούσε να βαρύνει μια υποχρέωση τον τομέα να έχει ένα ελάχιστο ποσό αποθηκευμένο ανα πάσα στιγμή, το οποίο θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει μόνο με το πράσινο φως ε, του κράτου. Και θα μπορούσε μάλιστα να έχει τοποθετηθεί ω σημείο αποθήκευση σε γειτονική χώρα. Αυτό συνδυάζεται μια χαρά με την περιφερειακή προσέγγιση που επιλέγει ο κανονισμό. Τώρα, για την τροφοδοσία. Όντω, είναι διαφορετικό από το κριτήριο της ε, ε, των υποδομών. Πρόκειται δηλαδή για διακοπή, για πρόβλημα τεχνικής φύσεως στον αγωγό. Ενώ η τροφοδοσία η αφορά όχι διακοπή, μάλλον ε, δεν αφορά πρόβλημα στις ε, υποδομές, στους αγωγούς ή αλλού. Είναι διαφορετική λοιπόν περίπτωση και ο ε, ε, καταναλωτή βεβαίω πρέπει να έχει τη δυνατότητα τροφοδοσία ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι υποχρέωση του παρόχου. Κατά την άποψή μου, αυτό σημαίνει ότι τον βαραίνει μια υποχρέωση που όμω πιστεύω ότι υπάρχει ήδη δυναμή τη οδηγία για την ε, αγορά φυσικού αερίου. Οπότε δεν είναι σαφές γιατί ο κανονισμό αυτό περιέχει σχετική διάταξη επίση. Και υπάρχουν και δύο πρότυπα διαφορετικά μεταξύ του με διαφορετικές προθεσμίες. Ηλεκτρική ενέργεια. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η αγορά φυσικού αερίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ του. Για το φυσικό αέριο πολλές φορές χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πολλές φορές μέχρι το 60% του συνόλου. Επιπλέον η ηλεκτρική ενέργεια με φυσικό αέριο είναι εναλλακτική λύση έναντι της αιωλικής ε, και ηλιακής ενέργεια. Και βεβαίω, ε, όπως το ηλεκτρικό χρειάζεται αέριο και το αέριο χρειάζεται ηλεκτρικό. Ε, καυστήρες ας πούμε δεν χρησιμοποιούνται πολλές φορές, δεν λειτουργούν χωρίς ηλεκτρικό. Ο κανονισμός ε, που έχουμε επιτάπτως δεν ρυθμίζει αυτό το θέμα. Δεν ρυθμίζει το θέμα δηλαδή τις ε, σχέσεις μεταξύ της ηλεκτρικής και ενέργειας και, της, του φυσικού αερίου. Η διασφάλιση των σταθερών τιμών δεν είναι ασφαλές, δεν είναι από μόνο του επαρκές μέτρο θα πρέπει να εξασφαλίζεται και η ε, προσκοπτή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για τις αντίστροφες ΡΕΣ. Η κρίση του ενεργείου του 2009 μας δίδαξε ότι το αέριο δεν μετακινείται εύκολα στην Ευρώπη ούτε, ανατολικά, ούτε από ανατολικά δυτικά, ούτε από βόρεια προ τα νότια. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο είχαμε προβλήματα με την επιστροφή τη ροή ή επειδή δεν υπήρχαν ισχυρέ σύμβασει που να το επιτρέπουν. Τώρα βεβαίω τα περισσότερα προβλήματα έχουν επιληθεί. Θα πρέπει όμω να γίνουν και περαιτέρω προσπάθειε, ίσονο θα έλεγα σημασία, όπω είπε και ο συνάδελφο, και υπάρχει και οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το πακέτο αναθέρμανση τη οικονομία. Το κατά παρελθόν δεν έγινε αυτό, γιατί ο οικονομισμό έλεγε ότι οι επενδύσει αυτέ ε, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τους χρήστες της χώρες. Ε, οι χρήστες όμως σε αυτές τις γειτονικέ χώρες επίσης ωφελούνται. Οπότε ο, ο διαμεσολαβητής ε, ε, μάλλον η αγορά το απέρριψε αυτό. Γι' αυτό με τον κανονισμό αυτό αλλάζει και είναι πολύ καλό. Βεβαίω ο οργανισμό ίσω να είναι υπερβολικό, ζητώντα όλου του διασυνδέσει να έχουν δυνατότητα αντιστροφή των ροών. Δύσκολα θα το πετύχουμε αυτό. Από την άλλη όμω, η αντιστροφή της ροής και η εφαρμοσιμότητα των διασυνδετών είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει εγγύηση όταν η αγορά από μόνη της δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Χρειάζεται μια αξιολόγηση του κανόνα N-1 πριν από την εφαρμογή αυτού του πρώτου και τελευταίου σημείου για τις οργανωτικές ικανότητες που έχουμε. Μια διαταραχή, μια διακοπή της παροχής φυσικού αερίου χρειάζεται άμεση δράση για την αποφυγή blackout αερίου blackout ε, αερίου είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να επανακάμψει πολύ εύκολα, αλλά για το φυσικό αέριο τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει οι τεχνικοί να επισκεφθούν όλα τα σπίτια για να διασφαλίσουν και να διαπιστώσουν να λειτουργεί σωστά. Κάθε χώρα λοιπόν θα πρέπει να προετοιμαστεί για τέτοιε διακοπέ παροχή φυσικού αερίου και θα πρέπει να έχει οργανωτικέ ικανότητε τέτοιε όπως ε, τεχνικές ασκήσεις, προσωμιώσεις, ένα εγχειρίδιο και οδηγίες που θα πρέπει να υποβάλει σε δοκιμασίες και με τις γειτονικές χώρες για να ξέρει ανά πάσα στιγμή ότι μπορεί το αέριο να κυκλοφορεί μεταξύ των χώρων. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο, το TSO για την ηλεκτρική ενέργεια θα πρέπει να συμμετάσχουν και αυτές, αυτές τις επίγουσες διαδικασίες. Αυτά ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ και για τις πληροφορίες και την αξιολόγηση της πρότασης. Επόμενος ομιλητής, Μάρσελ Κράμερ, είναι πρόεδρος της ε, Gas Infrastructure Uni. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ, πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση να σα αποτείνω το λόγο σήμερα το απόγευμα. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομο. Νομίζω διάφορε από τι απαραίτητε που είχα να ε, κάνω έγιναν ήδη από του προλαλήσαντε. Καταρχήν, είναι σαφέ, προφανώ ότι το φυσικό αέριο είναι σημαντικό συνεργαστής για την ε, ε, τροφοδότηση με ενέργεια. Και το φυσικό αέριο είναι το πιο καθαρό ορυκτό καύσιμο και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χρήση του στο μέλλον. Και γι' αυτό από δικά μας είναι λογικό και σημαντικό οι κυβερνήσεις να καθορίσουν ένα πλαίσιο που να προβλέπει το θέμα της ε, ανταγωνιστικότητα και ρευστότητα των αγορών φυσικού αερίου. Και εγώ θα αναφερθώ εδώ στη τρίτη δέσμη ε, που, του έργου που έχει επιτελεστεί για το θέμα αυτό και θα πρέπει να τονίσω ότι πολλά ακόμα θα πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η έγκαιρη εφαρμογή τη τρίτη δεσμή και θα πρέπει να σκεφτούμε τον συνδυασμό μεταξύ αυτών που συζητάμε σήμερα ε, εδώ και τις εφαρμογές της τρίτης δέσμης. Ε, εκτός από την ασφάλεια του εφοδιασμού είναι πάρα πολύ σημαντικό το πού και πώς θα πρέπει να ενδυναμωθεί. Γιατί οι επενδύσεις συνήθως κινητοποιούνται από την αγορά. Επενδύουν κάποιες εταιρείε γιατί οι... εκείνοι που και πως θα πρεπει να ενδυναμωθει γιατι οι επενδυσει συνηθως κινητοποιουνται απο την αγορα επενδυουν καποιες εταιρειε γιατι εκεινοι που προμηθευουν το αέριο και οι αγοραστές θέλουν το αέριο να πάει από το α στο β. Πολλέ φορέ αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται διακανονισμένο σύστημα. Οι ειδικοί όλοι μπορούν να οδηγήσουν σε αποφάσει ε, τη κυβέρνηση ότι πρέπει να υπάρχουν συμπληρωματικέ υποδομέ που δεν κινητοποιούνται από την αγορά. Και τότε τίθεται το θέμα πού θέλουμε τι τύπου συμπληρωματικέ υποδομέ για να εξασφαλίσουμε τον εφοδιασμό. Τι είναι αυτό που δεν μπορεί να λυθεί από την αγορά ή από τις υποδομές που υπάρχουν. Ο κ. Φανάιμεν αναφέρθηκε στο θέμα του κανόνα του νήμιον 1. Αυτό νομίζω ότι είναι χοντρικό ε, μέσο για να καταλήξουμε σε μια απάντηση για το πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, θα φτάσει το φυσικό αέριο έγκαιρα για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί αυτή η νέα υποδομή που δημιουργείται με το νήμιον 1. Και υπάρχει επίση το θέμα το ποιο θα πληρώσει. Πάντα σημαντικό. Ποιοι είναι οι σαφεί ε, χρηματοδοτικοί κανόνες που εξασφαλίζουν ένα ίσο και δίκαιο πεδίο παιδείας για όλους. Τέλος, πώς ενσωματώνεται η ισχύοντες κανονισμοί στην εφαρμογή της τρίτης δέσμης. Όλες οι διατάξεις επίσης που ισχύουν στα κράτη-μέλη και σε κοινοτικό επίπεδο πώς θα συμφορθούν. Θέλουμε βέβαια να αποφύγουμε περιττές επενδύσεις του δημοσίου χρήματος. Πιστεύουμε ότι αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με συνεχή έντονο διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων συγγνώμη, και των εταιριών. Και η GIE έχει τη δυνατότητα και τη βούληση να προχωρήσει προς την λόγω αυτή. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρο. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κράμερ, για την σύντομη και ακριβή σας αυτή παρουσίαση. Και έτσι θα έχουμε περισσότερο χρόνο για την ε, συζήτηση. Κατόπιν θα θέλω να δώσω το λόγο στον καθηγητή Δ. Μάρκο Ολίβερ Μπέτσιγκερ που είναι ε, διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου για την ε, Οικονομία της Ενέργειας στην Κολονία. Κύριε καθηγητά Μπέτσιγκερ, δική σας, ε, έχετε το λόγο. Χαίρομαι που είμαι εδώ και μπορώ να αναπτύξω κάποιες σκέψεις για δύο ζητήματα. Πρώτον, στην κολονία κάναμε μία ανάλυση της κρίσης του Ιανουαρίου και εδώ έχω κάποιες πρόσθετες πληροφορίες από αυτές που έδωσαν οι προλαλήσαντες και δεύτερον, τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης με βάση κάποιο μοντέλο μπορούν να μας οδηγήσουν σε κάποιες προτάσεις για τον κανονισμό. Όπως είπαμε λοιπόν, τον Ιανουάριο είχαμε μια διατάραξη της ροής από την Ουκρανία που είχε μετά ως αποτέλεσμα τις ε, σοβαρές αλλαγές στην κατεύθυνση ε, της ροής του αερίου στην Ευρώπη. Κανονικά το χειμώνα είναι η ροή από Ανατολή προς Δύση και το μοντέλο μας εδώ πέρα μας δείχνει βεβαίως την ε, ιδανική αντίδραση της, ε, του κλάδου σε αυτό το συμβάν μας δείχνει την ε, αλλαγή της κατεύθυνσης από τη Δύση προς την Ανατολή. Κάποια αποτελέσματα τώρα επιβεβαιώνουν αφενός αυτό το οποίο, αυτά τα οποία ακούστηκαν. Το μοντέλο μας δείχνει ξεκάθαρα πως ήταν ε, πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος των αποθεμάτων, ειδικά των γερμανικών και των ιταλικών και των ευρωπαϊκών βεβαίως. Και βλέπουμε εδώ πέρα δύο σημαντικά στοιχεία. Το μοντέλο ελάχιστου κόστους, ε, αποστολής με ελάχιστο κόστος μας δείχνει πως δεν θα ήταν δυνατόν να προμηθεύσουμε την Ανατολική Ευρώπη πλήρως με αέριο κατά τη διάρκεια της κρίσης, ακόμα και σε μια κατάσταση ελάχιστου ε, κόστους, οπότε ακόμα και με κεντρικό σχεδιασμό με βάση τους γεωγραφικούς περιορισμούς δεν θα μπορούσε να αποφύγει τις διαταραχές. Το μέγεθος των διαταραχών βεβαίως του μοντέλου δεν συγκρίνεται με τις πραγματικές διαταραχές γιατί δεν έχουμε πραγματικά δεδομένα αλλά βλέπουμε σαφώς πως είναι αναπόφευκτες οι διαταραχές ήταν αναπόφευκτες τον Ιανουάριο λόγω των περιορισμών του δικτύου. Το δεύτερο το οποίο μπορείτε να παρατηρήσετε είναι πως σε μια ιδεώδη αντίδραση ειδικά τα ιταλικά αποθέματα θα χρησιμοποιούνταν σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ε, κρίσης. Κάτι το οποίο βεβαίως ε, θέτει κάποια ερωτήματα για τη διαχείριση των ιταλικών αποθεμάτων. Υπολογίσαμε επίσης με το μοντέλο τον αντίκτυπο το, του οριακού κόστους ε, του να προμηθεύσουμε τις διάφορες περιοχές της Ευρώπης και εδώ πέρα βλέπετε την διαφορά στην τιμή λόγω της ε, διαταραχής αυτής και βλέπετε πως στα κόκκινα σημεία εκείνα ε, δεν θα είχαμε εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια της κρίσης και πράγματι εκεί είχαμε και διαταραχές ε, και στην πραγματικότητα. Επίσης, αυτό το οποίο δεν βλέπετε εδώ πέρα είναι πως οι διαφορές των τιμών που παρατηρήθηκαν στο γερμανικό κόμβο εμπορίας ανταποκρίνονται λίγο πολύ στην ανάλυση μας και βλέπουμε πως ολόκληρη η βόρειο Δυτική Ευρώπη έμεινε λίγο πολύ ανεπηρέαστη και το πρόβλημα ήταν στην Ανατολική Ευρώπη. Υπόθηκε ήδη πως ε, σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι αντιστροφές των ροών και δεν μπόρεσαν βεβαίως όλες οι υποδομές να το κάνουν αυτό, οπότε κάναμε για την ίδια περίοδο 40 ημερών άλλη μία προσωμείωση με την υπόθεση πως ε, όλοι οι αγωγοί μπορούν να κάνουν ε, αντίστροφες ροές. Και βλέπετε στη διαφάνεια πως ακόμα και αν είχαμε αντίστροφες ροές σε όλους ε, τους Αυγούστου θα ε, είχαμε και πάλι διατραχές με την κρίση αυτή που προέκυψε. Οπότε η αντιστροφή της ροής, η διπλή ροή, δεν λύνει εντελώς το πρόβλημα. Η πιο σημαντική διπλή ροή επί τη ευκαιρία είναι από την Τουρκία προς την Βουλγαρία. Αν πάω στην προηγούμενη διαφάνεια βλέπετε πως η, Βουλγαρία, η προμήθεια Βουλγαρίας και Ρουμανίας από τον Νότο μας βοηθάει στο να μειωθεί η έκταση του κόκκινου χρώματος στον χάρτη. Αναφέρθηκε πως ήταν κρίσιμος ο ρόλος ε, των αποθεμάτων και πως η Ευρώπη ήταν τυχερή Κατά κάποιον τρόπο αυτό το οποίο βλέπετε εδώ πέρα είναι τα αποθέματα διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών το χειμώνα του 2008 και το χειμώνα του 2009 μετά την κρίση και βλέπετε πως τον Απρίλιο του 2009 το επίπεδο των αποθεμάτων είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι ήταν στον Απρίλιο του 2008 με τον χειμώνα του 2008 και 2009 να έχει λίγο πολύ ίδιες ε, ε, μέσες ε, θερμοκρασίες. Οπότε έπεσαν τα αποθέματα πολύ περισσότερο από ότι το προηγούμενο έτος. Γιατί είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί υπήρχε ένα επιπλέον στοιχείο, η οικονομική κρίση στην Ευρώπη που οδήγησε σε μεγάλη μείωση της ζήτησης αερίου. Και εδώ πέρα προσωμείωσαμε το επίπεδο αποθεμάτων όπως θα ήταν εάν η ζήτηση του 0809 ήταν αυτή με του 0708 και ακόμα και με τις ίδιες θερμοκρασίες θα είχε εξαντληθεί το αέριο στο τέλος του Απριλίου και με αυτή την κρίση που είχαμε βλέπουμε πως μια παρατεταμένη κρίση ή ένας πιο κρύος χειμώνας το Φεβρουάριο και το Μάρτιο θα εξαντλούσε την ε, προσφορά και αν έχουμε ε, τον κίνδυνο ενός πιο κρύου χειμώνα έχουμε σοβαρά ζητήματα. Βεβαίως εδώ πέρα δεν έχουμε τις ε, απαντήσεις που θα είχαμε, τις αντιδράσεις που θα είχαμε σε περίπτωση ε, τέτοιες μεταβολής αγοράς από πλευράς προσφοράς και ζήτησης, αλλά βλέπετε πως ε, ε υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα της ε, κρίσης εδώ πέρα. Τώρα, ποια είναι τα μαθήματα από την ανάλυση αυτή με βάση το μοντέλο. Όπως σας είπα, το μοντέλο μας είναι ένας ιδανικός κόσμος και μετά το συγκρίνουμε με το τι συνέβη στην πραγματικότητα. Και βλέπουμε πως η αντίδραση του κλάδου είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό το οποίο βρήκαμε εμείς ως λύση ελάχιστου κόστους με κάποια ζητήματα υποδομής. Όπως σας είπα, είχαμε κάποια ζητήματα με τη χρησιμοποίηση των τελικών αποθεμάτων, αλλά Εκτός από αυτό, λίγο πολύ ε, ο κλάδος έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε με βάση τους περιορισμούς ε, των υποδομών. Αν ε, παρατηρήσουμε την αντίδραση του του κλάδου θα δούμε πως η συνεργασία ήταν κάπως ad hoc αλλά πολύ αποτελεσματική δεδομένων των περιορισμών των αντικειμενικών. Βλέπουμε λοιπόν πως υπάρχει μια αντίδραση ναι, έχουμε τέσσερα βασικά σημεία. Υπάρχουν σαφώς κάποια σημεία μποτιλιαρίσματος, αν θέλετε, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υποδομών. Εμφανίζονται λοιπόν κάποια σημεία που, που όταν υπάρχει κρίση δυσκολεύουν την ροή και δεν φαίνεται αυτό όταν λειτουργεί κανονικά η αγορά, οπότε πρέπει να ε, επιληθεί αυτό το ζήτημα. Νομίζω αναφέρθηκε και πριν αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Δεύτερον, βλέπουμε πως ήταν κρίσιμα τα επίπεδα των αποθεμάτων και δεν θα επαρκούσαν εάν ήταν πιο κρύος ο χειμώνα ή και εάν ήταν ψηλότερη η ζήτηση, δηλαδή αν δεν υπήρχε οικονομική κρίση ή και εαν ε, πήγαινε η κρίση πέρα από τις 40 ημέρες. Οπότε το επίπεδο των αποθεμάτων είναι κάτι που μας ανησυχεί. Τρίτον, υπήρχαν κάποια όρια στην διασυνοριακή αλληλεγγύη που ήταν σαφή. Ανέφερα το ζήτημα της Ιταλίας και της Σλοβακίας επίσης. Οπότε το τρίτο ζήτημα είναι η διασυνοριακή αλληλεγγύη. Πώς θα υπάρξει μια τέτοια αλληλεγγύη σε μια παρατεταμένη κρίση. Τέταρτον, υπάρχει μια... ένας ψηλός βαθμός πολυπλοκότητας στην διαχείριση των κρίσεων που δεν χρειάζεται και σημαίνει πως η γρήγορη αντίδραση σε περίπτωση κρίσης είναι δύσκολη. Λύθηκε ad hoc μέσω συνεργασία εταιριών και ρυθμιστικών αρχών. Καλό θα ήταν να είναι σαφείς οι κανόνες για περίπτωση κρίσης, ίσως με το να χαλαρώσουν ε, κάποιοι περιορισμοί που υπάρχουν για τις εταιρείε. Με βάση λοιπόν αυτά τα μαθήματα που ατλήσαμε από την κρίση θα θέλαμε να κάνουμε κάποια σχόλια στην ε, πρόταση αυτή που έχουμε τώρα μπροστά μας. Προφανώς με βάση την ανάλυση μας θέλουμε να έχουμε μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Η αρχή της επικουρικότητας ε, σωστά έχει τυποποιηθεί εδώ πέρα για περίπτωση Επίση Επίσης η τυποποίηση και εναρμόνιση και συντονισμό είναι επωφελή. Επίση θεωρούμε πως υπάρχει κάποιο περιθώριο βελτίωσης ειδικά στις εξή πτυχέ. Πρώτον, η κρίση κατέδειξε πως η αγορά και οι ανταγωνιστικές εταιρείες αντέδρασαν στα συμβάντα πάρα πολύ γρήγορα. Οι δυσκολίες κυρίως οφείλονταν ε, στην καθυστέρηση του να οργανωθεί η μεταφορά, οπότε νομίζουμε πως οι τιμές είναι ο καλύτερος τρόπος ε, για να διαμορφωθεί η χρήση του αερίου εκεί που χρειάζεται περισσότερο. Οπότε τα σχέδια εκτέκτου ανάγκης, εάν είναι πάρα πολύ τυποποιημένα και δεν έχουν ελαστικότητα, θα έχουν αντίστοιχο αποτέλεσμα, θα εμποδίζουν την ε, αποτελεσματική αντίδραση της αγοράς. Η ευελιξία ήταν κλειδί ευελιξία που επιδείχθηκε από όλου. Οπότε αν είναι πάρα πολύ άκαμπτα τα σχέδια εκτέκτου ανάγκη, θα ε, έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Δεύτερον, δεν είμαστε πεπισμένοι πως ε, σε μια κρίση μια παρέμβαση κρατών ή της Κομισιόν θα οδηγήσει σε αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς. Θεωρούμε πως η κατανομή των όγκων θα πρέπει να οργανώνεται κυρίως μέσω τιμών και της ε, λειτουργίας ανταγωνιστικών αγορών. Κατόπιν, όπως είπαμε, κατά την άποψή μας δεν θεωρούμε πως είναι οικονομικά αποτελεσματική η γενική ε, ροή ε, δύο κατευθύνσεων. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο παντού, οπότε δεν χρειάζεται να γίνουν και άχρηστες, μη απαραίτητες επενδύσεις. Και τέλος το κριτήριο νη 1 δεν φαίνεται πως επαρκεί για να εγγυηθούμε την ε, ασφάλεια ε, προμήθειας. Για να δούμε και το τι έγινε και τον Ιανουάριο. Το κριτήριο αυτό από μόνο του δεν επαρκεί και ίσως να είναι και λανθασμένο. Οπότε αυτά τα οποία καταδείξει το μοντέλο, χώρες οι οποίες καταδείξει το μοντέλο ότι είναι ασφαλείς, με τον ύπλην 1 δεν είναι ασφαλής. Έχουμε λοιπόν κάποιες προτάσεις για να βελτιωθεί η πρόταση αυτή, χωρίς βεβαίως να είναι πλήρης η αξιολόγηση. Πρώτα απ' όλα προτείνουμε να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ του ανταγωνιστικού τμήματος αγοράς και του ρυθμισμένου τμήματος αγοράς. Για το ανταγωνιστικό τμήμα της αγοράς θεωρούμε πως πρέπει να εμπιστευόμαστε τους μηχανισμούς αγοράς ακόμα και σε περίπτωση κρίσης. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να παρέμουν τα κράτη-μέλη και να χρησιμοποιήσουν την πολιτική ισχύ ή ακόμα και δικαιώματα ή ιδιοκτησιακά που έχουν σε εταιρείε για να προωθήσουν εθνικούς στόχους ε, εις βάρος της ευρωπαϊκής αλληλεγγύη. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος κατά την άποψή μας στον ε, ανταγωνιστικό τομέα. Όπως σας είπα, δεν θεωρούμε πως η καλύτερη λύση είναι άμεση παρέμβαση της Κομισιόν. Θεωρούμε πως καλύτερο θα ήταν ευθυγραμμισμένοι με άλλους ε, κλάδους αγοράς να υπάρξει τιμωρία ex post εκ των υστέρων. Για τον δε ρυθμισμένο τομέα της αγοράς ε, θεωρούν πως πρέπει να υποστηρίζει λειτουργία των αγορών ακόμα και σε περίπτωση κρίσης. Οπότε η τυποποίηση και η εναρμόνιση της νέας αγοράς βεβαίως στο μέτρο του δυνατού και μετά να είναι απλοποιημένες οι διαδικασίες για όλες τις εταιρείες τις εμπλεκόμενες κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Τρίτον, προτείνουμε τον ή πλην 1 να αντικατασταθεί από, ένα, ε, από μια προσέγγιση που θα βασίζεται σε συστήματα που θα ελέγχουν το, το βάρος που υπάρχει στο σύστημα γιατί αν επικεντρωνόμαστε μόνο στο νημιον 1 επικεντρωνόμαστε μόνο σε κάποιες μεγάλες ε, χώρες, ενώ θα πρέπει να δούμε και την ε, εικόνα και στις 27 χώρες. Τέλος, άποψή μας είναι πως πρέπει να δώσουμε βάρος στις υποδομές και όχι στις διαδικασίες. Οι διαδικασίες βοηθάνε, αλλά ποτέ δεν επαρκούν ασφάλεια εφοδιασμού θα έχουμε εάν εξετάσουμε τις υποδομές και τους όγκους, τις ποσότητες, δηλαδή πρέπει να ε, δείτε και να δώσετε κίνητρα στις κατάλληλες επενδύσεις, πρέπει να υπάρχει δηλαδή κάποια δυναμικότητα η οποία θα ε, περισσεύει ανά πάσα στιγμή και αυτό πρέπει να γίνει από ευρωπαϊκή σκοπιά δεύτερον τα επίπεδα αποθεμάτων είναι σημαντικά οπότε πρέπει να οριστούν να παρακολουθούνται και να υπάρχει άμεση συνεισφορά στα αποθέματα όπως επεσήμαναν και οι προηγούμενοι μιλητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες τώρα. Θα πρέπει τώρα να μοιράσουμε το χρόνο έτσι, ούτως ώστε όλοι όσοι θέλουν να υποβάλουν ερωτήσει να μπορέσουν να τις υποβάλουν. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Βίταλ Κφάντρας και μετά παρακαλώ ζητήστε το λόγο να γραφτεί το κατάλογο. Παρακαλώ. Yes, uh, thank you very much, Mr. Ευχαριστώ. Με την ιδιότητά μου του εισηγητού θα προσπαθήσω αργότερα να εξαγάγω κάποια συμπεράσματα. Τώρα, εις το παρόν στάδιο, το πρώτο που θα ήθελα να πράξω είναι να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες στην ακρόαση και να τους πω ότι είναι έτοιμοι να θητεύσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί έκαναν αυτό που εμείς καθημερινά κάνουμε. Δηλαδή, συμπίκνωσαν τον λόγο τους σε λίγων λεπτών σοφία. Πέραν τούτο θα ήθελα να πω ότι είναι άκρος από ικανοποιητικό για τα μέλη αυτά τη Επιτροπή, ότι όλα τα σημεία τα οποία αναφέρατε, με τον τρόπο μάλιστα που τα αναφέρατε, σαφώς συμμορφούνται και με τις δικές μας ανησυχίες και επιθυμίες και απόψεις. Και αυτό είναι πολύ καλό για μας. Γιατί ορισμένε φορές τις ακροάσεις ακούμε πράγματα, πώς να το πω, που απομακρύνονται πολύ από αυτά τα οποία εμείς αρχικώς πιστεύαμε. Όχι. Δεν ισχύει σήμερα αυτό. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και αυτό μας καθησυχάζει απόλυτα. Δύο είναι τα σημεία που θα ήθελα να θίξω και επί των οποίων θα σας παρακαλούσα ευγενώς να σχολιάσετε περαιτέρω η έννοια του προστατευόμενου πελάτου. Δεν μπήκε κανένας από σας σε λεπτομέρειες, αγαπητοί εμπειρογνώμονες, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε περισσότερα. Το δεύτερο, παρά το ότι όλοι σας, παρά το ότι όλοι σας, παρά το ότι όλοι σας αναφέρατε έναν σαφή, σαφή σκεπτικισμό, κάνατε κάποιες επικρίσεις για τον κανόνα N-1 θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας πιο λεπτομερώς από αυτού. Να μας κάνετε μια πιο, πιο λεπτομερή ανάλυση των τεχνικών, πρακτικών δυσκολιών του προτύπου του κανόνος της προσεγγίσεως θα έλεγα N-1. Σας ευχαριστώ. Προτείνω να συλλέξουμε τώρα κάποιες ε, παρατηρήσεις. Η κυρία Γαμπάλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ομιλητές για τις ε, πολύ πλήρεις και ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους. Συμφωνώ με τον τελευταίο μιλητή ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις υποδομές και πώς θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τα πλεονάσματα που χρειάζονται. Υπάρχουν θέματα λοιπόν που τίθενται. Χρειαζόμαστε διαφοροποίηση των υποδομών και διαφοροποίηση της τροφοδοσίας. Για να το πράξουμε αυτό γιατί δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στην πρόσβαση στον Ατλαντικό και να στραφούμε σε χώρες πηγής όπως οι χώρες της Δυτικής Αφρικής και να έχουμε πιο πολλές εγκαταστάσεις υγραερίου στην Ευρώπη. Δεύτερο οι απαιτούμενε επενδύσεις. Είναι πρόβλημα κοινό για όλους αλλά και για άλλους τομείς, όχι μόνο για το φυσικό αέριο και για την καθαρή ενέργεια και για την ασφάλεια τροφοδοσίας χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις στην Ευρώπη. Ανέφερε κάποιος ομιλητή το πακέτο αναθέρμανσης της οικονομίας αλλά και κάποια εγχειρίδια προς τους χρήστες δεν επαρκούν αυτά κατά την άποψή μου. Η κάλυψη της χώρας, η διασύνδεση με την Ισπανία και την Αλγερία έχουν απορροφήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των όσων δικαιούμαστε δυνάμει των διαρθρωτικών ταμείων. Άλλαξαν όμως οι καιροί και τώρα με την οικονομική κρίση θα πρέπει να σκεφτούμε πώς στο μέλλον θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε, θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις περαιτέρω προσπάθειε που πρέπει να κάνουμε για τις υποδομές στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κ. Φόμποντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα ω κοιόδη συζητητή των Σοσιαλδημοκρατών να συμφωνήσω με όσα είπε ο κύριο ε, εισηγητή. Πολύ συγκεκριμένε προτάσει. Έχω τρει ε, παρατηρήσει. Καταρχήν αναφέρομαι σε αυτό που είπε και ο κύριο Βίταλ Κβάτρο. Τι γίνεται με τον λεγόμενο προστατευόμενο καταναλωτή. Ε, η Κομισιόν αφήνει ανοιχτό κατά πόσον κάποιε περιφέρειες μπορούν να διευρύνουν την έννοια αυτή περισσότερο. Ρωτώ λοιπόν κατά γνώμη θα πρέπει να είναι στενή η έννοια του όρου αυτού και να ισχύει για όλη την Ευρώπη ενιαία ή θα μπορέσει κάθε κράτος μέλος ελεύθερα να αναφέρεται σε αυτή την έννοια μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ. Και όπως είπε και κάποιος ε, τι γίνεται και όσον αφορά την, ε, τους οικονομικούς λόγους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεύτερον, το θέμα των αποθεμάτων φυσικού αερίου όπως είπε και η Πορτογαλίδα συνάδελφος, θα πρέπει να συζητούν με το LNG. Γιατί καμιά φορά περισσότερες δυνατότητες LNG αντικαταστούν την εναγκαιότητα αποθεμάτων φυσικού αερίου. Και αυτό με το αναφέρθηκε ο κύριος Κράμερ, ο κύριος Σμέλτσερ κυρίως, ε, ανέφερε στο θέμα αυτό κατά πόσον βάσει του κανονισμού αυτού θα πρέπει να ε, αναφερθεί υποχρέωση για αποθέματα φυσικού αερίου η διεύρυνση των δυνατοτήτων υπήρχαν διάφορες ε, απόψεις επί του θέματος του παρελθόν και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι η ποσότητα των αποθηκευμένων ποσοτήτων σε διάφορες χώρες ε, μέλη είναι πολύ διαφορετικές για τεχνικούς λόγους, οικονομικούς, πολιτικούς είναι ενδιαφέρον ε, και εγώ από την Αυστρία, όπως και εσείς ξέρετε, έχουμε πολύ υψηλά επίπεδα υποθεμάτων, αλλά στην Ευρώπη τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Το τελευταίο ερώτημα αναφέρεται σε κάτι που δεν εθίγει. Το θέμα της ενημέρωσης ε, των εταιριών φυσικού αερίου προς την Κομισιόν. Αυτό δεν αναφέρεται καθόλου, αλλά αναφέρεται ότι υπάρχουν ε, απόρριτα τμήματα των ε, συμβάσεων που δεν θα πρέπει να μεταβιβαστούν. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Σμέλτσερ, οι διακανονιστέ τι κάνουν, έχουν τι απαραίτητε ε, ε πληροφορίε, τι γίνεται με το απόρριτο. Μήπω πάνω στο θέμα αυτό τη προώθηση ε, των πληροφοριών από την, ε, τη βιομηχανία παραγωγή φυσικού αερίου, θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε κάτι σχετικό. Ευχαριστώ. Επόμενο ήταν ο Έχω δύο ερωτήματα. Το ένα είναι γενικό απευθύνεται προς ε, ολόκληρο το πάνελ. Είναι τι ξέρουμε για τις ε, πιθανές οικονομικές συνέπειες ε, του κανονισμού, ειδικά όταν θα εισαχθεί το νη μείον Δεδομένων ε, των προθεσμιών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κανονισμό, τι γίνεται με τα βραχυπρόθεσμα προγράμματα επενδύσεων της, ε, του κλάδου. Υπάρχουν σχετικά σχέδια. Και δεύτερον, ε, προς τον κύριο Μπέτσουγκε, είπατε πως στην τελευταία κρίση υπήρχαν περιορισμοί στην διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Μπορείτε να μας εξηγήσετε την αιτία. Ήταν οικονομικοί περιορισμοί, ήταν πολιτικοί λόγοι ή υπήρχαν τεχνικά ζητήματα. Εάν συμφωνείτε θα ακούσουμε ακόμη έναν συνάδελφο τον κύριο Πάσκα Ευχαριστώ. Εις ό,τι αφορά τα συμβάντα του Ιανουαρίου του 2009, η Σλοβακία επλήγει σε πολύ μεγάλο βαθμό από την κρίση και θα πρέπει να πω ότι η Σλοβακική Δημοκρατία έχει τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου από κατανάλωσης δεν θα έπρεπε κανονικά να έχει προκύψει πρόβλημα. Ακόμα και σε καιρό κρίσης θα έπρεπε το κράτος να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Και όμως δεν είχαμε θέρμανση. Και όμως πέρασαν τρεις εβδομάδες με πάυση των δραστηριοτήτων των βιομηχανιών. Γιατί, διότι το αέριο είναι στα χέρια δυτικοευρωπαϊκών συμφερόντων. Και η χώρα μου υπέγραψε μια συμφωνία δυνάμει της οποίας το αέριο έπρεπε να περνάει από την Τσεχία και ίσως στο μέλλον δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρει μόνο το που βρίσκεται η αποθήκη ή το αποθηκευμένο αέριο, αλλά οι σχέσεις των Ευρωπαίων και των Ευρωπαϊκών κρατών μεταξύ τους. Αυτό είναι το ζητούμενο κυρίες και κύριοι. Αλλιώς οι ιδιοκτήτες των αποθεμάτων δεν θα δώσουν πολλές φορές τη δυνατότητα απελευθέρωσης αυτού του αποθηκευμένου φυσικού αερίου, ακόμα και εκεί που το χρειάζεται ο τόπιος πληθυσμός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν ακόμα πάρα πολλές ζητήσει το λόγο δεν ξέρω που θα αντέξουν οι εμπειρογνώμονες να έχουμε και κάποιες συμπληρωματικές ερωτήσεις και μετά να απαντήσετε. Παρακαλώ, κύριε Μπουτιχόφερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες για τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας έδωσαν. Και θέλω να θέσω δύο ερωτήματα. Το ένα ερώτημα σχετίζεται με Μία παρατήρηση του καθηγητού κυρίου Μπετσίουγε. Αναφερθήκατε σε έλλειψη διαμεθορικής ελληνικής. Cross-border solidarity. Δεν θα σας παρακαλέσω να το διευκρινίσετε κάπως καλύτερα αυτό που είπατε, ιδίως σε σχέση και με το εξή θέμα. Ποια είναι η ευθύνη πρόληψης των επιμέρους των μελών σε σχέση με την ελεγγύη προς άλλα κράτη-μέλη. Πώς εξισορροπούμε δηλαδή αυτές τις δύο ιδέες. Υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια που μπορούν να ξεφύγουν από τα σημερινά πολιτικά προβλήματα. Και το δεύτερο ερώτημα προς τον κύριο Σμέλτσερ και προς τον καθηγητή κύριο Μπετσούγερ. Αναφερθήκατε και άλλοι πραγματικές στην αναγκαιότητα συμπληρωματικών υποδομ... επενδύσεων συγγνώμη στις υποδομές. Αυτό που δεν έφερε κανένας όμως είναι κατά πόσο ενδεχομένω επενδύσεις στην μείωση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου, δηλαδή επενδύσεις για υψηλότερη αποτελεσματικότητα της χρήσης του φυσικού αερίου, θα πρέπει να είναι οικονομικά πιο ενδιαφέρουσα από τις επενδύσεις σε συμπληρωματικές υποδανειμές. Ίσως υπάρχει κάποιο σημείο τομής μεταξύ των δύο αυτών. και θα μπορούσαμε ε, μέσα στα πλαίσια μια ορθολογική ε, συνολική στρατηγική για την, ε, τον θεσμό του ΕΛΟΥ να το λάβουμε υπόψη μα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Θα ήθελα να δώσω στου προγνώμενου τώρα τη δυνατότητα σύντομα να απαντήσουν. Ο κ. Σμέλτσερ καταρχήν. Μάλιστα, θα ήθελα να αρχίσω με το θέμα του ορισμού του προστατευόμενου πελάτη ή καταναλωτή. Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να είναι σαφής ο ορισμός μέσα στο πλαίσιο του κανονισμού και να μην ε, προβλέπει πολλούς ε, περιορισμούς και θα πρέπει να εφαρμοστεί αυστηρά γιατί θα πρέπει ακριβώς να λάβουμε υπόψη ότι ακριβώς μεγάλοι καταναλωτές, βιομηχανικοί δηλαδή καταναλωτές, έχουν τη δυνατότητα υποκαταστάτων. Και ακριβώς αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη στην ε, ασφάλεια του εφοδιασμού. Γι' αυτό αυτή η έννοια του προστατευόμενου πελάτη θα πρέπει να είναι ενιαία και ε, να εφαρμόζεται περιοριστικά. Δεύτερον, το οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, το θέμα της υποχρέωσης ε, στην ε, πρόσβαση στα αποθέματα ή την υποχρεωτική τήρηση αποθεμάτων. Έχω να πω ότι εδώ τα διάφορα κράτη-μέλη ε, έχουν πολύ διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος ε, και δεν υπάρχουν παντού αποθέματα. Στις χώρες όπου δεν υπάρχουν ή υπάρχουν ανεπαρκή αποθέματα μπορεί να υπάρξει τελικά ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κινούμεται και σε μια απελευθερωμένη αγορά όπου ενδεχόμενο ε, η αποθήκευση για μια χώρα να γίνεται στη γειτονική χώρα. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η αποθήκευση θα πρέπει να γίνεται κάτω από προθέσεις αγοράς και θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι χρειαζόμαστε αδιαφανή πρόσβαση στα αποθέματα αυτά με γνωστούς όρους συμβολέων για να μπορούν όλοι να έχουν τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσουν. Περαιτέρω ερώτημα αφορούσε στο θέμα της ε, εποπτείας ε, της ε, ασφάλειας εφοδιασμού. Αυτό εξαρτάται από την κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε από τη χρησιμοποίηση του φυσικού αερίου. Εμείς δηλαδή σαν αρχή για να το αξιολογήσουμε χρειαζόμαστε μια σαφή νομική βάση να συλλέγουμε αυτά τα στοιχεία. Παραδείγματος χάρη ποια είναι και η ευελιξία η συμβατική που υπάρχει, δηλαδή όλα τα συμβόλαια αυτά έχουν μία ευελιξία 10-15% και είναι σημαντικό ποιε είναι οι συμπληρωματικέ ποσότητε που θα μπορούσαν να έχουν, ποιε είναι οι εναλλακτικέ δυνατότητε αγορά φυσικού αερίου. Αυτό όλα τα χρειάζονται οι αρχέ για να μπορέσουν να τιμήσουν κατά πόσον η κατάσταση μπορεί να επιληθεί με όρου αγορά ή αν θα πρέπει να υιοθετηθούν ε, μέτρα κρίσης, που είναι βέβαια πάντα η τελευταία διόδοση. Και ίσως για το πρότυπο νήμιον 1. Πιστεύουμε ότι αυτό το πρότυπο μπορεί να έχει αποτελέσματα ε, και βλέπουμε ότι ιδίω στον τομέα της ε, αντίστροφης ροής οι επενδύσεις δεν είναι τεράστιες Πολλές φορές είναι μικρές οι επενδύσεις αυτές, όπου το κύριο πρόβλημα είναι η κατανομή του κόστους. Και όσον αφορά το πρότυπο νήμιον 1, θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει σαφής υποδιέρεση σε πρότυπα υποδομής για να μπορέσουν έτσι οι έμποροι να αγοράσουν τα, τις που χρειάζονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να αναφερθώ σε λίγα μόνο σημεία καθώς ε, πιστεύω πως το τέλος θα καλυφθούν όλα. Πρώτο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι το εγκροποιημένο φυσικό αέριο και η αγορά της λεκάνης του Ατλαντικού, όπως ε, λέγεται στην αγορά, που συμπεριλαμβάνει και τη Δυτική Αφρική. Υπάρχουν πολλά έργα που υλοποιούνται. Αυτή τη στιγμή ο κλάδος ε, κοιτά να δει πώς θα διαφοροποιηθεί η προμήθεια μέσω terminals ε, επαναεριοποίησης όπως λέγονται. Υπάρχουν πάρα πολλά έργα στην ακτή του Ατλαντικού, επέκταση στο Βέλγιο, νέο έργο στο Ρότερνταμ και πολλά έργα στη Μεσόγειο. Οπότε γίνεται πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο. Η ανησυχία μέχρι πρόσφατα ήταν πως ε, καλά είναι τα... η καταστάση υποδοχής αλλά από πού θα έρθει το υγροποιημένο αέριο. Βλέπουμε πως αλλάζει όμως η εικόνα, η διαθεσιμότητα πρόθεσμα. φαίνεται πως θα εξαρτηθεί και από τις λεγόμενες μη συμβατικές πηγές αερίων στη ΣΥΠΑ και υπάρχει κάποια δυνατότητα για τέτοια παραγωγή και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Και το ζήτημα είναι αν μπορούν να τα βρουν εταιρείε και κυβερνήσεις για να εκμεταλλευτούν αυτούς τους πόρους παραγωγικά και υπεύθυνα. Νομίζω πως αυτές οι συζητήσεις για το μη συμβατικό αέριο θα αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία και είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Οπότε, ο συνδυασμός περισσότερων ε, τερματικών σταθμών, ε, ίσως και κάποιας καλύτερης διαθεσιμότητας λόγω της παγκόσμιας αγοράς και των μη συμβατικών πηγών αερίου θα μειώσει την ε, ευαισθησία μας σε διαταραχές ε, της ε, παροχής καθώς και στην διασύνδεση με τους υπάρχοντες αγούς. Θίξατε το ζήτημα των επενδύσεων. Η εμπειρία μας είναι πράγματι πως οι επενδύσεις είναι κρίσιμο ζήτημα ε, δεν γίνεται ευκολότερο για προφανείς λόγους αλλά θεωρούμε πως σε γενικές γραμμές ε, με πολλές εταιρείες και επενδυτικά ταμεία κοιτάνε σοβαρά τις επενδύσεις. Το βασικό ερώτημα είναι η απόδοση της επένδυσής μου αναλογή με τον κίνδυνο τον οποίο διατρέχω. Ε, και ειδικά όταν είναι να φτιάξουμε μια διασυνοριακή σύνδεση θα αποδώσει επένδυσή μου και στις δύο πλευρές των σύνορων και δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις οποίες αυτό είναι εξαιρετικά αμφίβολο και πρέπει να γίνει δουλειά. Και γνωρίζω πως η νέα αριθμιστική αρχή ακριβώς θα επικεντρωθεί στα δύο συνοριακά ζητήματα έτσι ώστε όταν έχουμε δύο συνοριακές ε, επενδύσεις να είναι αυτές αποτελεσματικές και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Ε, μπορώ να φέρω αρκετές περιπτώσεις στις οποίες αυτό δεν γίνεται αυτή τη ε, στιγμή και υπάρχουν αντιδράσεις μεταξύ εθνικών συστημάτων για καθαρά ιστορικούς λόγους. Αυτό πρέπει να το δούμε, να συνεργαστούμε και ξέρω πως το Κοινοβούλιο κάνει μεγάλη προσπάθεια. Για τα αποθέματα τώρα υπάρχουν πολλές σχετικές πρωτοβουλίες, πολλά έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βεβαίως είναι και ζήτημα υπεδάφους από γεωλογικούς όρους καθάρα δεν είναι κάθε υπέδαφος κατάλληλο για αποθήκευση φυσικού αερίου Και βεβαίως το ζήτημα είναι εάν υπάρχουν και χρήστες διατεθειμένοι να υπογράψουν συμβάσεις για να ξεκινήσει και το έργο με καλές προοπτικές και αν υπάρχουν και εταιρείε διατεθειμένες να επενδύσουν σε σχέση με τις άλλες εναλλακτικές που έχουν. Αυτό δεν σημαίνει πως αυτομάτως θα πρέπει να οδηγηθούμε σε υποχρεωτικά αποθέματα, αν και νομίζω πως ε, πρέπει να γίνει μια ανάλυση για να δούμε πού πραγματικά υπάρχει έλλειψη στο κάθε σενάριο. Συμφωνώ με τον κύριο από την κολονία που ανέφερε διαφορετικά σενάρια. Ίσως σε κάποια κατάσταση όταν μιλάμε για την κορύφωση της ζήτησης μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Δημόσιο Ταμείο κάποιο είδους ε, αποθήκευση. Τέλος, για τα, τις οικονομικές επιπτώσεις του νήμιον 1. Είναι και αυτό ένα σενάριο, αλλά μπορούμε να πούμε πως εάν χρησιμοποιήσουμε ένα τόσο αμβλή μέσο, μπορεί να φτάσει το κόστος τα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Και τέλος, ναι, η αποτελεσματική χρήση ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντική και εμείς ως υποδομών υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης του φυσικού αερίου. Μειώνει το κόστος και μειώνει βεβαίω και το πόσο εκτεθειμένοι είμαστε. Και πρέπει να καταβάλουμε κάθε σχετική προσπάθεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριο Μπόιν. Και εγώ να απαντήσω σε ορισμένα από τα ερωτήματα που θέθησαν. Ποιοι είναι οι προστατευόμενοι πελάτες. Ποιοι είναι. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσουν οι πολιτικοί. ποιους θέλουν να προστατεύουν από τις διαταραχές και τις κρίσεις. Πάντως από τεχνικής απόψεως ως προστατευόμενος πελάτης θεωρείται ως ο ή οσδήποτε που δεν μπορεί να εξασφαλίσει την τροφοδεσία του μόνος του. ο μέσος καταναλωτής ουσιαστικά Ο εισηγητής είπε ότι εμείς ασκούμε κάποια επίκριση στον κανόνα N-1. Όχι εγώ πάντως. Έθεσα κάποια ερωτηματικά για το πώς διατυπώνεται στον κανονισμό, αλλά γενικά το κριτήριο του N-1 μια χώρα, μια περιοχή θα πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους διαταραχές όχι της τροφοδοσίας αλλά των υποδομών του είναι καλό πράγμα. Τώρα βέβαια θα πρέπει να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Τι είναι λογικό και τι όχι. Ας πούμε η αγωγή, η αραγωγή να πηγαίνουν στα σημεία αποθήκευσης, ε, υγροποίηση του αερίου, όχι. Πάντως, ως αρχή, είναι πολύ σωστή. Για την αποθήκευση, όπως είπε ο κύριος Κράμερ, είναι πολλές οι τρέχουσες πρωτοβουλίες. δεν είναι η εμπορική πτυχή των πραγμάτων που χωλένε. Όχι. Γι' αυτό και πιστεύω ότι δεν είναι δυνατή η υποχρεωτική επιβολή της αποθήκευσης σε όλες τις χώρες τουλάχιστον, γιατί δεν είναι σαφές ακόμα πώς αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό οι διάφορες χώρες. Για υποχρεωτικά μέτρα θα πρέπει να έχουμε μια ad hoc προσέγγιση αναχώρα ή αναπεριοχή. Για ορισμένους θα μπορούσε η υποχρεωτική αποθήκευση να είναι μια λύση. Για την Ουγγαρία ας πούμε όπως είδε το αποφάσι η Ιταλία. Αλλά δεν είναι unisex αυτή η λύση. για το υγροποιημένο αέριο υπάρχουν πολλές τέτοιου είδου υποδομές αναφέρθησαν και το νούμερο βασίλειο ας πούμε έχει μεγάλες ε, ικανότητες στον τομέα μπορεί και με τη διασύνδεση να βελτιωθεί η κατάσταση Υπάρχει και θέμα έκθεσης όμως στην παγκόσμια αγορά. Οι διασυνδέσει είναι περιφερειακό ζήτημα. Και όταν υπάρχουν διαταραχές είναι το ευάλωτο σημείο του συστήματος. Ενώ το LNG είναι πολύ πιο ευάλωτο. Σε ό,τι φορά τι πηγές δηλαδή τροφοδοσία. Όσο έχουν τα πράγματα τώρα υπάρχουν πολλές ε, ε, μονάδες υγροποίησης στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική. προ το παρόν λοιπόν δεν είναι πρόβλημα, αλλά για το μέλλον ε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε όλοι τσμήματα μιας παγκόσμιας αγοράς. Όπως και για το πετρέλαιο που άρχισε να μετακινείται κάποια στιγμή παγκόσμια με τα δεξαμενόπλια. Το ίδιο κάποια στιγμή θα μπορούσε να γίνει και με το φυσικό αέριο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις οικονομικές συνέπειες, ή τις δημοσιονομικές συνέπειες του κανονισμού. Εδώ σαν ήδη κάποια παραδείγματα, κάποια αριθματικά στοιχεία, ας πούμε η αντίστροφη ροή, πώς συγκρίνεται με την οικονομική ζημία. Οποιοςδήποτε κανονισμός ε, εφαρμοστεί, στόχο έχει την πρόληψη οικονομικών ζημιών για το κράτος και τις διαταραχές τροφοθήσεις για τα νοικοκυριά. Οπότε είναι θέμα το πώς θα ασφαλιστούν αυτές οι επενδύσεις κατά του ενδεχομένου να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Νομίζω ότι έτσι απαντώ στα ερωτήματα που μου ετέθησαν. Ευχαριστώ. καθηγητής ο κύριος ευχαριστώ. Θα απαντήσω πρώτα απ' όλα τις ερωτήσεις που απευθύνθηκαν σε μένα και μετά θα κάνω και κάποια σχόλια σε αυτά τα οποία είπαν οι άλλοι ομιλητές για την διασυνοριακή αλληλεγγύη να διευκρινίσω. Από όσο ξέρω δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις έλλειψης αυτής της αλληλεγγύης. Το μοντέλο μας όμως έχει κάποιες ενδείξεις ε, που εγείρουν κάποια ερωτήματα, ειδικά όσον αφορά τα Ιταλικά αποθέματα και το τι συνέβη επίση και με τη Σλοβακία στο τέλος της κρίσης. Οι παρατηρήσεις μας αυτές ανταποκρίνονται και στα στοιχεία που προέκυψαν και στον τύπο και μιλώντας με τους ανθρώπους του κλάδου. Δεν υπάρχουν όμως αποδείξεις. Είναι σημαντικό όμως το ζήτημα αυτό να το δούμε όταν μιλάμε για τέτοια ρύθμιση και για να το δούμε σαφώς καλό είναι να έχουμε τυποποιημένα κριτήρια εναρμονισμένα και στις 27 χώρες για το τι επίπεδα ασφάλειας ε, της προμήθειας πρέπει να έχουμε και βεβαίως αυτό σχετίζεται και με το πώς θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τα επίπεδα αποθεμάτων. Εάν είμαστε μέσα του χειμώνα τον Ιανουάριο πρέπει να ληφθεί μία απόφαση πόσο μέρος των αποθεμάτων αποδεσμεύουμε και πόσο κρατάμε για το Φεβρουάριο και το Μάρτιο. Οπότε ένα εναρμονισμένο κριτήριο θα ήταν ε, πολύ θετικό και για να έχουμε βεβαίως και εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να είναι ευρωπαϊκό. Γιατί μεταφέρεται το αέριο από την μία χώρα στην άλλη, στην εσωτερική αγορά. Το δεύτερο ερώτημα που αφορούσε εμένα ειδικά ήταν το ζήτημα της αποτελεσματικής χρήσης και της ζήτησης του αερίου και είναι πολύ σωστό ερώτημα. Η ανάλυση που σας ε, έδειξα και τα κριτήρια που προτείνει η Κομισιόν χρησιμοποιούν τα τωρινά δεδομένα της ζήτησης για να αξιολογήσει την ασφάλεια νη μείον ή ένα σενάριο για τον Ιανουάριο με βάση τα δεδομένα του Ιανουαρίου. Και προφανώς βεβαίως, η επενδύσεις στις υποδομές χρειάζονται χρόνο και κατά τη διάρκεια αυτών των επενδύσεων μπορεί η ζήτηση να αυξηθεί π.χ. για την παραγωγή ενέργειας αλλά μπορεί και να μειωθεί λόγω της αποτελεσματικότερης κρίσης στα νοικοκυριά που αναφέρατε. Οπότε για να αξιολογηθεί η ασφάλεια της παροχής πρέπει να κοιτάμε σε έναν ορίζοντα δεκαετίας και για να έχουμε μια σταθερότητα βεβαίως σε βάθος δεκαετίας και από εκεί θα προκύψουν και οι επενδυτικές αποφάσεις. Νομίζω αυτό, το, αυτό είναι το ζήτημα που εξετάζει και η Ένωση των ε, Ρυθμιστικών Αρχών αυτή τη στιγμή σε κάποια πιο γενικά ζητήματα τώρα. Πρώτα απ' όλα το κριτήριο νήμιον 1. Δεν θα ήθελα τώρα να ακουστεί ότι είπα εγώ ότι δεν είναι χρήσιμο. Όχι, είναι καλό, αλλά δεν επαρκεί. Δεν ενσωματώνει πλήρως μια ευρωπαϊκή ε, οπτική και την σχέση μεταξύ των διαφόρων ε, χωρών. Οπότε πρέπει αυτό να συμπληρωθεί με μια ευρωπαϊκή και συστημική οπτική. Δεύτερον, και αναφέρθηκε αυτό, ε, παραλείπει το ζήτημα των όγκων των ποσοτήτων που είναι σημαντικό και για, τις, ε, για τα αποθέματα και υπάρχει βεβαίως και κάποιο περιθώριο ερμηνείας που κάτι το οποίο δεν ε, μας βοηθά ιδιαίτερα για το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Ένα σχόλιο ακόμα συμφωνώ πλήρως με την αξιολόγηση πως ε, αυξάνεται βεβαίω η ασφάλεια ε, όσο έχουμε περισσότερες τέτοιες δυνατότητες και αν έχουμε και τέρμιναλ βεβαίως ε, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται υπό κανονικές συνθήκες αλλά μόνο σε καιρούς κρίσης ποιος θα πληρώσει γι' αυτά. Επίσης να επισημάνω πως ε, το υγροποιημένο φυσικό αέριο δεν είναι η μόνη υποδομή που βελτιώνει την ασφάλεια παροχής. Παραδείγματο χάρη η επένδυση Nord Stream με μια σύνδεση βορρά-νότου θα αυξήσει τον όγκο που μπορεί να μεταφερθεί στην Ανατολική Ευρώπη από μια διαφορετική πορεία εάν διαταραχθεί πάλι η διαδρομή μέσω Ουκρανίας. Οπότε βλέπετε πως ε, οι υποδομές ε, αγωγών είναι εξίσου χρήσιμες με το LNG. Το ίδιο ισχύει και για τον Αμπούκο μέσω της Μεσογείου. Μετά υπήρχε το ζήτημα για το επίπεδα των αποθεμάτων και αν θα έπρεπε ήδη εδώ πέρα να οριστεί μια σχετική υποχρέωση. Η προσωπική μου άποψη είναι η εξής θα πρότεινα πως σαφώς πρέπει να αποτελέσει τμήμα της πρότασης το να οριστούν τα πρότυπα των κατάλληλων επιπέδων και να υπάρχει επιτήρηση των προτύπων αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να, να συμπεριληφθούν και διατάξεις για το τι θα πρέπει να γίνει όταν, εάν φτάσει η Ευρώπη στο συμπέρασμα πως ε, δεν ανταποκρίνονται πλέον τα επίπεδα αυτά στα κριτήρια που έχουμε. Δεν νομίζω πως αυτή τη στιγμή πρέπει να εξετάσουμε άμεσες ε, συνεισφορές σε στρατηγικά αποθέματα αλλά πρέπει να είναι σαφές ε, το τι θα γίνει αν η Ευρώπη θεωρεί πως δεν υπάρχουν επαρκή αποθέματα. Και τέλος, να επαναλάβω ένα σχόλιο που έκανα. Είχαμε το ερώτημα για τις ε, πληροφορίες, ε, τις επίμαχες αυτές πληροφορίες ε, που θα πρέπει ο κλάδος να δίνει στην Κομισιόν. Όπως ερμηνεύω εγώ την πρόταση αυτή και την διάταξη αυτή, νομίζω πως αυτό κυρίως στοχεύει στην πιθανή έλλειψη διασυνοριακής αλληλεγγύης. Βεβαίως αυτό μπορεί να συμβεί αν π.χ. ανταγωνιστικές εταιρείες στα κράτη-μέλη επηρεάζονται από τους πολιτικούς και δεν ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις τιμές. Κάτι το οποίο βεβαίως θα είναι αρνητικό για τον κλάδο είναι να συμβεί. Οπότε ναι, πρέπει να έχουμε μια τέτοια διάταξη. Η άποψή μου είναι πως ε, μια διάταξη που θα προβλέπει άμεση παρέμβαση της Κομισιόν είναι πάρα πολύ δυνατός ε, μηχανισμός. Εγώ θα προτιμούσα μια κύρωση εκ των υστέρων εάν δεν συμμορφώνονται στις τιμές οι εταιρείες. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Τώρα έχουμε πίεση χρόνου. Κολεάν αποσιάζει. Τσουκαλάς. Αν είναι δυνατόν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να πληροφορηθώ σε ποιο ποσοστό το LNG, είτε για καθημερινή τροφοδοσία είτε σε περιπτώσεις κρίσεως, αποτελεί ε, πηγή λύσεων γιατί εμείς ε, μπορέσαμε να βοηθήσουμε την φίλη Βουλγαρία κατά την περίοδο της κρίσης από τον σταθμό της Ραβδιθούσας με τα LNG. Άκουσα την παρατήρηση για τις διαφοροποιημένες υποδομές. Καταλαβαίνω ότι η παγκόσμια, η παγκόσμια ναυτιλία έχει όλα και όλα 300 πλοία μεταφοράς ε, αερίου. Υπάρχει περίπτωση να θεωρηθούν η ναυπήγηση, η επιδότηση κατασκευής πλοίων μεταφοράς αερίου σε ένα σενάριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα χρησιμοποιεί LNG μια, ε, μια πιθανότητα. Τέλος θα ήθελα να ξέρω μήπως με τα σχέδια των νέων αγωγών προωθούμε όπως είναι ο Ναμπούκο. Εκείνο που κάνουμε είναι να αντικαταστήσουμε μια εξάρτηση όπως είναι η ρωσική εξάρτηση αέριου δηλαδή μέσω της Ουκρανίας αντικαθιστούμε με μια εξάρτηση που δεν είναι τόσο καλύτερη όπως είναι το αζέρικο ιρανικό αέριο μέσω της Τουρκίας. Και τέλος μόνο ότι στις είδα στις παρουσιάσεις την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από, το, από τα φυσικά αποθέματα της Αιγύπτου ή της Λιβύης για το 2030 μου διαφεύγει αν υπάρχει όχι πολιτική επάνω σε αυτό και θα ήθελα να την πληροφορηθώ. pane eh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ pouze. Ήθελα να σας πω ότι πραγματικά ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί στην τελευταία κρίση του φυσικού αερίου γιατί υπήρχαν διάφορα θετικά για μας. Βέβαια την επόμενη φορά δεν σημαίνει ότι θα συντρέχουν ε, τα ίδια θετικά σενάρια. Έχω κάποιες παρατηρήσεις για τον Ήμιον 1. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπεσέ τι γίνεται όσον αφορά αυτές τις δοκιμασίες κρίσης που ενδεχομένως αντικαταστήσουν τον Ήμιον 1. Και επίσης προς όλους του εμπειρογνώμονε, θα ήθελα να υποβάλω την ερώτηση τη χρηματοδότηση των μέτρων αυτών. Ε, θεωρείτε ότι είναι καλό εταιρείε ε, όταν οι, τα πράγματα πάνε καλά έχουν κέρδη και όταν πρέπει να δημιουργήσουν δίκτυα και να απτύξουν δυναμικό κλπ που θα είναι κατάλληλα για να απορροφήσουν και παρεκκλήσεις της αγοράς. Στην περίπτωση αυτή λέω είναι σωστό να ζητούν ε, χρήματα φερρυπίν από τα εθνικά ταμεία ή τα ευρωπαϊκά ταμεία. Αυτό είναι ηθικό. Και επίσης θα να ρωτήσω ε, το στρατηγικό πρόβλημα που θα πρέπει να επιληθεί δηλαδή να συνδεθούμε καλύτερα με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Είναι σωστό. Ευχαριστώ και Σκάλες. Thank Ευχαριστώ. Από τις ε, πρώτες διαφάνειες εδώ πέρα διαβάζω λέτε πως η λειτουργία της αγοράς είναι η καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια ε, παροχής. Μετά από αυτό το οποίο είπε ο κύριος ε, Μπόλτς. Διαφάνεια ε, ακόμα και σε καιρούς ε, κρίσης. Ωραία πράγματα. Βεβαίως για να υπάρχει ένας μηχανισμός αγοράς πρέπει να υπάρχει μια αγορά που λειτουργεί και για να λειτουργεί η αγορά πρέπει το αέριο από τη μία άκρη της Ευρώπης, από ένα σημείο στην Ευρώπη να μπορεί να πάει σε ένα άλλο. Στην πρώτη παρουσίαση είχαμε μια τιμή, κάτι το ευχαριστώ, 80 με 90 εκατομμύρια ευρώ, αλλά βλέπετε πως για την Ανατολική Ευρώπη το λέτε, κάτι το οποίο συμφέρει σε σχέση με τις ζημίες του περασμένου χειμώνα. Οπότε, μετά από όλο αυτό το συνειρμό Μπορείτε να μας πείτε πόσο κοστίζει να συνδέσουμε τα διάφορα τμήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη για να λειτουργεί όλη αυτή η αγορά, γιατί βεβαίως ε, η αντίστροφη ροή λειτουργεί στους ε, υπάρχοντες αγωγούς. Τι γίνεται για τα κομμάτια εκείνα της Ευρώπης που είναι αποκομμένα από τα υπόλοιπα. Συμφωνώ, ναι, να λειτουργούν οι αγορές, αλλά πρέπει να υπάρχει υποδομή. Και ποιο είναι το κόστος. Ευχαριστώ, Charles Chichester. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Μπρεζίνας ήδη απήντησε σε ένα, μάλλον εξήγησε ένα ερώτημα γιατί ζήτησε από τον καθηγητή Πετσούγκη να εξηγήσει περαιτέρω στοιχεία, να δώσει περαιτέρω στοιχεία εις ό,τι αφορά τις δοκιμές. Ε, το ε, και εγώ αυτό το ερώτημα. Τώρα, για τον κύριο Βαμπόμεν, που αν τον κατάλαβα καλά, είπε ότι δεν είναι υπέρ του ορίου των 60 ημερών. Γιατί? Μπορείτε να μας πείτε. Στο κάτω-κάτω μιλάμε για μια επίγουσα κατάσταση. Δεν μιλάμε για μια συστηματική ή μια διαρθρωτική έλλειψη. 60 μέρες για μια επίγουσα περίπτωση είναι αρκετές. Αν δεν βρούμε λύση σε 60 μέρες, ε, τότε πότε θα τη βρούμε. Διότι μετά τις 60 μέρες γίνεται διαρθρωτικό το πρόβλημα. Μου έχουν πει δε ότι μία απώλεια του 10% είναι χαμηλή για να δικαιολογείται η λήψη αποφάσεων επιγόντων μέτρων. Δεν δική μου άποψη. Σας, ερωτώ, να, σας ζητώ να μου πείτε τη δική σας. Και η τελευταία μου ερώτηση, Κράμερ. Έχετε επίγνωση των τελευταίων δημοσιευμάτων, τα οποία διάβασα εγώ, ότι υπάρχει πολύ περισσότερο φυσικό αέριο από αυτό το οποίο υποθέτουμε ότι υπάρχει λόγω των αλλαγών στην αγορά αυξημένη αποτελεσματικότητα, τροφοδοσία υγραερίου έχει αυξηθεί όλα αυτά δεν μας καθιστούν λιγότερο εξαρτημένους από εισαγωγές εξανατολών ή μήπω αυτό είναι έτσι ένας βραχυπρόθεσμος ε, μια βραχυπρόθεσμη αισιοδοξία ή μήπω αντίθετα σηματοδοτεί κατά την άποψή σας μια πιο μακροπρόθεσμη ε, διαφορά στην αγορά. Κυρία Φόρντ, ευχαριστώ πολύ. Το ερώτημα μου αφορά την ασφάλεια. των εγκαταστάσεων αποθήκευσης του φυσικού αερίου. Στη δικιά μου περιφέρεια, το 2005 τεράστια έκρηξη σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου. Η μεγαλύτερη στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν είχε γίνει οποιαδήποτε άλλη στιγμή έγινε 4 ώρα το πρωί μια Κυριακή αν είχε γίνει, επαναλαμβάνω, οποιαδήποτε άλλη μέρα και οποιαδήποτε σχεδόν άλλη ώρα θα είχαμε ε, πολλές απώλειες ζωής. Γι' αυτό οι κάτοικοι της περιοχής μου ανησυχούν ιδιαίτερα για το θέμα της ασφάλειας ή ασδήποτε εγκατάστασης αποθήκευσης. Στην περιφερειά μου Υπάρχουν κάποιες πολύ, μια, πολύ, κάποιες πολύ παλιές εγκαταστάσεις της δεκαετίας του 60 σε ένα μικρό νησάκι 45.000 κατοίκους και ένα δρόμο μόνο. Οπότε χάρηκα πολύ με αυτά που είπατε για τα πρότυπα, τα υψηλά πρότυπα αποθήκευσης, συντήρηση κτλ. Γιατί είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ. Ποιες είναι οι απόψεις σας ημών ως εμπειρογνώμονες χωρίς να λέμε καλό το μέτρο αλλά όχι εδώ, αλλού. Τι μπορούμε να κάνουμε για την ασφάλεια των πολιτών μας ε, στα πλαίσια αυτά. Ευχαριστώ. Κύριος Μέρκος, τελευταίος ομιλητής. Uh, uh, Κυρία Μέρκος. Uh, Ευχαριστώ. Υποστηρίζω το ερώτημα του κ. Τσίτσεστερ και εγώ το ίδιο ήθελα να ρωτήσω πάνω κάτω. Στις κάτω χώρες θεωρούμε ότι είναι θέμα που αφορά την ίδια την εικόνα της κοινότητας. Τι, πώς ορίζεται η κρίση και πότε προκύπτει. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη όλων των εμπειρογνωμόνων. Εξ όσων γνωρίζω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει το 10% της ε, συνολικής ε, τροφοδοσίας ενέργεια. Εμείς έχουμε ως ελάχιστο στις κατοχώρες 20%. Άρα ποια είναι η άποψή σας. Ευχαριστώ. Θα δώσουν οι προγνώμες τώρα σύντομες απαντήσεις παρακαλώ. Ένα-δύο λεπτά. Ο καθένα να συγκεντρώσει την προσοχή στις ερωτήσει που του υπευλήθησαν. Να μην πάρουμε τρει-τέσσερι ε, απαντήσει για κάθε ερώτηση. Ο κ. Σμέρτσερ. Äh, θα ήθελα να αρχίσω με το θέμα της χρηματοδότησης των επενδύσεων υποδομών που έχουν σε στόχο την ε, ασφάλεια της ε, ε, τροφοδότησης και του φωτισμού. Αυτό ή θα είναι μια επένδυση η οποία μπορεί να περάσει στην αγορά, δηλαδή δυναμικό μεταφορών που έχει κάποια ζήτηση και εκεί γίνεται βέβαια η επένδυση Ένα τμήμα των επενδύσεων της αντίστροφης ροής επίσης μπορεί να χρηματοδοτηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θα μπορούν να υπάρξουν ε, ε, πελάτες που θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και επενδύσεις ε, που έχουν μόνο σε στόχο την περίπτωση κρίσης και θεωρούμε ότι αυτό το κόστος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο κόστος δικτύου που βέβαια θα πρέπει να αναγνωριστεί μέσω του διακανονισμού. Ε, εδώ αναφερόμαστε και στην περίπτωση στην οποία οι επενδύσεις είναι προ και άλλων χωρών και εκεί θα πρέπει να γίνει κάποια κατανομή του κόστους. Και σχετικά δεν πρέπει να ξεχνάμε το θέμα του ότι το κόστος ε, του δικτύου είναι περίπου το 5-7% ε, του συνολικού κόστους. Δηλαδή ακόμα και διπλασιασμός του κόστους δεν θα είχε τις ίδιες επιπτώσεις όπως η αύξηση της τιμής του αερίου. Αυτό έτσι για να έχετε κάποιο συσχετισμό κατά νου. Όσον αφορά τώρα τον ορισμό της κρίσης, ε, σύμφωνα τις εμπειρίες που έχουμε εμείς, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κρίση στην οποία ε, μία σαλοπός μπορεί να αντιμετωπιστεί με μέτρα της αγοράς. Και αυτό θα πρέπει να κρυθεί μέσα στα πλαίσια της εποπτείας της κρίσης. Αυτός ο ορισμός ε, έχει και σαν στόχο να επιτρέπεται κάτω το δυνατόν ο διακανονισμός από την αγορά. Και γι' αυτό λέμε ότι κρίση είναι μετά από το σημείο με το, μέχρι το οποίο μπορεί να κανονιστεί η αγορά μόνη της. Όσον αφορά την ανάπτυξη για άλλα δίκτυα, αναφέρθηκε ο εγωγός Ναμπούκο. Εγώ εμεί θεωρούμε ότι υπάρχει ένα πλεονέκτημα, υπάρχουν εναλλακτικέ δυνατότητες μεταφοράς. Αν δούμε την ζήτηση φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ιδίως λόγω της ζήτησης για μονάς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, καλό είναι να έχουμε όλες τις δυνατότητες κατά νου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, το LNG. Αναφέρθηκε το θέμα της Βουλγαρίας. Εγώ δυστυχώς δεν έχω ε, στα χέρια μου κάποια περαιτέρω μελέτη για να δώσω συγκεκριμένες απαντήσεις. Αλλά θα ήθελα να τονίσω κάποια γενικά θέματα σχετικά με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, μια εγκατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα των στενοπών. Ναι, είναι καλό για αυτό το λόγο να υπάρχουν δερματικές μονάδες LNG. Αλλά τώρα πώς θα τροφοδηθεί αυτή η δερματική μονάδα είναι σημαντικό θέμα επίσης. Πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Κατά δεύτερον, στην περίπτωση αυτή μπορεί να υπάρχει συμφωνία με τον πολιτή όσον αφορά την τιμή, ούτως ώστε να είναι ανταγωνιστική. Γιατί όπως ελέγχθη προηγουμένως, λόγω της ανάπτυξης της αγοράς του LNG υπάρχει αυτή η κατάσταση κατά την οποία ε, ε, προωθούνται τα οι ροές αυτές στις αγορές τις οποίες ε, έχουν το μεγαλύτερο κέρδος. Πώς μπορούμε λοιπόν να έχουμε μια εγγύηση ασφάλειας γιατί ακόμα και αν υπάρχει θέμα δεν μπορεί κανένας να πληρώσει την ε, υπερυψωμένη τιμή. Επίσης το θέμα της των tankers ε, δεν είναι προβληματικό αυτή τη στιγμή για το LNG. Δεν υπάρχει στενοπόση εκεί και δεν νομίζω ότι χρειάζεται εκεί να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να γιατί θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο μπορεί να υπάρχει τερματικό σταθμό, κατά πόσο μπορεί να υπάρχει προμήθεια με, σε μια τιμή επαρκή και βέβαια αυτό ο τερματικό σταθμό θα πρέπει να συνδέεται κάπω με το δίκτυο. Και το θέμα είναι υπάρχει δυνατότητα αυτή ούτως ώστε να υπάρχει αποτελεσματική επένδυση και σε αυτό το τομέα. Μετά, η χρηματοδότηση. Ποιος πληρώνει, πώς πληρώνει. Εγώ δεν μπορώ παρά να σας παρουσιάσω τα παραδείγματα που είδα μέχρι στιγμής για αυτού του τύπου μέτρων κρίσης, όπως σε πολλές χώρες Ένα παράδειγμα είναι βέβαια τα αποθέματα πετρελαίου. Δεν υπάρχει απόλυτα παραλυσμός μεταξύ των δύο βέβαια, γιατί πρόκειται για διαφορετικά καύσιμα. Αλλά υπάρχει, λέω, για το πετρέλαιο κάποιος διακανονισμός σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση αποφασίζει ποιο είναι το ελάχιστο επίπεδο που χρειάζεται και εάν η βιομηχανία δεν μπορεί να προσφέρει το επίπεδο αυτό γίνεται κάποια προσπάθεια ούτως ώστε το αρχικό κόστος να κατανεμηθεί σε όλη την αγορά. Και έτσι τα ποσά που πληρώνουν οι μεμονωμένοι καταναλωτές ή οι εταιρείε είναι ελάχιστα. Ε, τέθη το θέμα για τα πρόσφατες δηλώσεις του τύπου ότι υπάρχει περισσότερο αέριο στη διάθεση κλπ. Αυτό διαβάζει κανένας που και που Βέβαια, οι ε, λόγω οικονομική κύκλοι προσπαθούν να βρουν περισσότερα κοιτάσματα αερίου και πετρελαίου. Εγώ αναφέρθηκα στο μη συμβατικό αέριο στις ΗΠΑ και βοηθιέται έτσι ο εφοδιασμός στη χώρα αυτή και το LNG τώρα που δεν πάει στη ΣΥΠΑ πάει αλλού βέβαια. Αυτό λοιπόν βοηθάει και τους άλλους. Αλλά βέβαια θα πρέπει να δούμε ποιε είναι αυτές οι δυνατότητες και στην ευρωπαϊκή αγορά. Και τέλος, το θέμα που τίθεται είναι κατά πόσον η Ευρώπη είναι διεθνώς ανταγωνιστική για, σαν ε, στόχος εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Ε, ανταγωνιστική λέω όχι μόνο όσον αφορά την τιμή, αλλά κατά πόσον μπορεί έγκαιρα να δημιουργήσει τι υποδομέ που χρειάζονται για να μπορέσει το αέριο αυτό να περάσει πραγματικά στου καταναλωτέ. Αυτό είναι η τρίτη δέσμη. Άμεση. Υπάρχουν τα σχετικά πλαίσια σε όλα τα κρατημέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να κατασκευαστεί η υποδομή που χρειάζεται. Η οικονομική ε, κύκλοι θα θέλουν βέβαια να κάνουν τις επενδύσεις αυτές ε, βασιζόμενες σε φυσικούς, ε, φυσιολογικούς όρους οικονομικούς. Υπάρχουν πολλοί που θέλουν να επενδύσουν εφόσον θα υπάρχει κάποιο, ε, κάποια δυνατότητα χρησιμοποίηση και κέρδους μέσω της υποδομής αυτής. Και τέλος συμφωνώ απόλυτα με την προειδοποίηση που νομίζω ότι άκουσα όσον αφορά το θέμα της οικονομικής κρίσης που δείξει σε λιγότερη ε, ζήτηση. Όλοι οι δείκτες αυτή τη στιγμή ε, τείνουν να δείχνουν υψηλότερη ανάγκη μεταφορών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καλό λοιπόν να χρησιμοποιούνται οι πόροι που υπάρχουν εκτός νοσής και να υπάρχει σχετική υποδομή. Το θέμα της αποθήκευσης του φυσικού αερίου πραγματικά είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Ε, το θέμα της ασφάλειας μέχρι στιγμής ε, τα αποτελέσματα ήταν πάρα πάρα πολύ θετικά. Άρα πρέπει να είμαστε πάντα σίγουροι ότι επενδύουμε στις υποδομές αυτές όπως πρέπει, να επαγρυπνούμε και να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν νέες ε, γνώσεις και παραδείγματο χάρη με τα νέα αυτά τερματικά για το LNG θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις γνώσεις που έχουμε για τις εγκαταστάσεις για να είναι απόλυτα ασφαλής και είναι σημαντικό οι εθνικές ε, αρχές να συμβάλλουν με την εμπειρία τους και ό,τι μπορεί να γίνει προς την κατεύθυνση αυτή είναι θετικό. Τέλος, όσον αφορά τον ορισμό της κρίσης, συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Το κλειδί είναι ότι όταν μιλάμε για τη διαχείριση της κρίσης θα πρέπει καταρχήν να είμαστε σίγουροι ότι τα τρέχοντα σχέδια για τις υποδομές, για τα δίκτυα, για το LNG και για την αποθήκευση εξακολουθούν να πραγματοποιούνται. Να έχουμε το σωστό περιβάλλον γι' αυτό, ούτως ώστε αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πολύ επιλεκτικά μετά να δούμε ποιος θα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των αρχών και των ενδιαφερομένων οικονομικών κύκλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ να είμαστε σύντομοι γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα ε, χρόνου. Κύριε Ε, σύντομα λοιπόν. Βουλγαρία. Νομίζω πράγματι βοηθήθηκε η Βουλγαρία από Πνευσικό αέριο που ήρθε μέσω Ελλάδος. Απλά δεν υπήρχαν συμβάσεις για να περάσει τη Βουλγαρία και χρειάστηκαν κανένα δύο εβδομάδες. Το όριο των 60 ημερών για το αν είμαι υπέρ ή κατά. Κάνω μία διάκριση όπως και ο κανονισμός μεταξύ του προτύπου υποδομών και παροχής το πρότυπο υποδομών είναι εάν είναι, εάν είναι σε θέση η υποδομή να παραδώσει το αέριο ακόμα και αν υπάρχουν μεγάλες βλάβες. Ανεξαρτήτως του αν υπάρχει αέριο. Τώρα, για τις υποδομές, γιατί 60 ημέρες. Πάντα δεν θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ακόμα και αν ε, έχει πάθει βλάβη το μεγαλύτερο κομμάτι. Τώρα, για το πρότυπο της παροχής, φαντάζομαι πως θέλουμε να καλύψουμε ορισμένες ημέρες ε, από την διακοπή παροχής από μια πηγή. Τώρα, το όριο της ε, εκτάκτου ανάγκης, εγώ δεν θα ήμουν υπέρ κανενός ορίου. Οι κυβερνήσεις και οι κομισιόν πρέπει να παρακολουθούν την αγορά από κοντά. Συνήθως οι αγορές αντιμετωπίζουν τις διακοπές, είναι συνηθισμένες μόνο εάν υπάρχει απόδειξη πως η αγορά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα συμβάν, έχει φτάσει η στιγμή για να παρέμβει η Κομισιόν ή το κράτος. Το να υπάρχει ένα προκαθορισμένο όριο μπορεί να προκαλέσει κερδοσκοπία από την αγορά για το εάν έχουμε φτάσει ή όχι αυτό το όριο, αν θα παρέμβει το κράτος ή όχι. Ας ε, αφήσουμε τη λειτουργία της αγοράς στην αγορά καλύτερα. Για την ασφάλεια νομίζω ο κύριος Κράμερ ήδη είπε πολλά την ασφάλεια από ατυχήματα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως ε, πλην του LNG τα περισσότερα σημεία αποθήκευση είναι εξαντλημένα πεδία φυσικού αερίου. Δηλαδή προϋπήρχε εκεί φυσικό αέριο και αποθηκεύεται ξανά για την παροχή φυσικού αερίου τώρα, αν θα υπάρχει επάρκεια στο μέλλον. Τις τελευταίες, την τελευταία δεκαετία ανακαλύπτουμε περισσότερο φυσικό αέριο από όσο χρησιμοποιούμε, οπότε προστίθεται συνεχώς. Ε, μιλάμε σε παγκόσμια κλίμακα. Δυστυχώς στην Ευρώπη εξαντλούνται αποθέματα. Σας ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μπετσούγκε. Κάποια σχόλια για το τεστ αυτό αντοχής. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει δύο στοιχεία. Πρώτα απ' όλα ένα λεπτομερές μοντέλο ροής ε, του αερίου συμπεριλαμβανομένων και των αποθεμάτων των πραγματικών αυτή τη στιγμή και τέλος ελάχιστες προδιαγραφές παροχής για το, για το κάθε είδος καταναλωτή για ακραίες θερμοκρασίες τις ερχόμενες εβδομάδες. Εάν μπει αυτό στο μοντέλο και μετά γίνει μια ανάλυση νη πλην ένα στις, στην Ευρώπη των 27 μπορούμε να υπολογίσουμε τις ημέρες μέχρι την ε, διαταραχή. Βεβαίως σε αυτή την περίπτωση το νη 1 δεν πρέπει να το δούμε μόνο ατομικά ε, για να δει εδώ, αλλά πρέπει να δούμε τουλάχιστον σε επίπεδο χώρας. Ε, δηλαδή, εάν στην κάθε χώρα σταματήσει η εισαγωγή, χρησιμοποιώντας διάφορες ε, πηγές, μάλλον θεωρώντας ότι έχει διακοπεί από διάφορες πηγές και όχι μόνο να θεωρήσουμε ότι έχει κοπεί η παροχή από έναν μόνο αγωγό, μπορούμε να υπολογίσουμε μετά σε πόσες μέρες θα έχουμε διακοπή και ποια θα είναι η πρώτη χώρα που θα πληγεί. Και μετά βεβαίως εάν θέλουμε να δούμε πόσες μέρες θέλουμε να επιζήσουμε από αυτές τις συνθήκες έχουμε το αποτέλεσμα που επιζητούμε. Βεβαίως σημαντικό εδώ πέρα είναι και το ευρωπαϊκό μοντέλο ροής αερίου που είναι η αφετηρία. Δεύτερον για τη χρηματοδότηση θεωρώ πως τελικά θα πρέπει να το πληρώσουν οι πελάτες του δικτύου. Και αν είναι να το πληρώσουν αυτό πρέπει να δούμε και πώς οι ρυθμιστικές αρχές θα αντιμετωπίσουν τις επενδυτικές προτάσεις για κάποιες ε, περιτές ε, δυναμικότητες. Κάτι βεβαίως το οποίο θα πρέπει να δουν και οι ρυθμιστικέ αρχές για το πώς δεν πρέπει να οδηγηθούμε σε υπερβολέ. τέλο. αυτό το οποίο και ο κ. Κράμερ για την μακροπρόθεσμη εξέλιξη. Βραχυπρόθεσμα βλέπουμε πως υπάρχει ένα πλεόνασμα LNG στη λεκάνη του Βορειοατλαντικού. Μακροπρόθεσμα τα μοντέλα μας δείχνουν πως ναι, το υγροποιημένο φυσικό αέριο θα αυξηθεί δραματικά παγκοσμίω, αλλά για την Ευρώπη μέσω μακροπρόθεσμα το αέριο από τους αγωγούς από την γειτονιά της Ευρώπης ε, θα είναι ανταγωνιστικό για την Ήπειρό μας. Δύο παρατηρήσεις για να κλείσω. Μία για το ζήτημα της ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην ποιότητα των εγκαταστάσεων αυτών ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη που οφείλονται κυρίως στην γεωλογία και άρα δεν μπορούν να αλλάξουν. Οπότε εδώ πέρα είναι σαφές ότι χρειάζεται μια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Και μπορούμε εδώ πέρα να έχουμε θετικά αποτελέσματα από την ε, συνέργεια, καθώς μπορεί να αυξηθεί η ασφάλεια παροχής με χαμηλότερο κόστος ε, σε περίπτωση κρίσης. Δηλαδή να αποθηκευτεί το αέριο στις χώρες που έχουν την καλύτερη γεωλογία γι' αυτό. Και τέλος αναφέρθηκε πως ο Ναμπούκο παραδείγματο χάρη θα αυξήσει την εξάρτησή μας από χώρες διέλευσης όπως Τουρκία. Μία παρατήρηση για την Τουρκία. Όπως ε, προκύπτει από την ανάλυση, η κατεύθυνση διπλής ροής Βουλγαρίας-Τουρκίας θα βοηθούσαν πάρα πολύ στο να βοηθήσουν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία σε περίπτωση κρίσης. Αλλά αυτό το οποίο δείχνει η ανάλυση φαίνεται στη διαφάνεια είναι πως η αντίστροφη ροή από την Τουρκία στην Βουλγαρία σε περίπτωση κρίσης αυξάνει το κόστος για την Τουρκία. Οπότε από πλευράς αλληλεγγύης η αλληλεγγύη κοστίζει για την ε, Τουρκία και το ζήτημα είναι πώς θα διασφαλίσουμε ότι η Τουρκία θα είναι διατεθειμένη να επιδείξει αυτή την αλληλεγγύη σε καιρούς κρίσης και να διαθέσει τα πετούμενα κονδύλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμπεριγνώμενες εγκαρδιότατα. Να σας ζητήσω συγγνώμη που κάπως σας πιέσαμε λόγω έλλειψης χρόνου προς το τέλος. Τρία πράγματα ακόμα. Η Κομισιόν θέλει κάτι να πει σήμερα ή μπορούμε να το αναβάλουμε. Κύριε Πενουά, θέλετε κάτι να πείτε τώρα. Τώρα, εντάξει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που οργάνωσε αυτή την ακρόαση άκρος ενδιαφέρουσα Συμφωνούμε και στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο πρέπει να προχωρήσουμε με αυτό το σχέδιο κανονισμού κανείς από όσο άκουσα εγώ τουλάχιστον δεν αμφισβητεί την αρχή που διέπει το κείμενο Είπανε όλοι ότι θα πρέπει να το βελτιώσουμε. Και βεβαίως δεν είναι εύκολα θέματα αυτά, αλλά είναι σαφές ότι είμαστε διτεθειμένοι να το πράξουμε. Υπάρχουν και πολύ χρήσιμες ιδέες επιτάπητος από αυτό. Οι υποδομές ε, και η τροφοδοσία είναι τα δύο πιο βασικά στοιχεία και τα αντίστοιχα πρότυπά τους. Πρώτα απ' όλα για να να κατανοήσουμε καλύτερα το περιεχόμενο του προτινομένου κανονισμού ε, και για να διευκρινίσουμε διάφορες έννοιες που χρησιμοποιούνται. Δηλαδή δεν είναι απόλυτα εύληπτη αυτή η φόρμουλα του νήμιον 1. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν και θα διευκρινιστούν. Ο κύριος Πετσούγκε ανέφερε σαφώς ότι δεν έχουμε τις απαραίτητες υποδομές για να διασφαλίσουμε την ε, αγαστή λειτουργία της αγοράς. Δεν είχαμε τον Ιανουάριο του 2009. 1,4 δις ευρώ δίδονται για τη χρηματοδότηση αυτών των διασυνδέσεων που δεν είχαμε τον Ιανουάριο αλλά και για τη χρηματοδότηση του reverse flow της αντίστροφης ροής. Είναι και αυτό κάτι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στα πλαίσια αυτής της συζήτησης. Επίσης ε, βεβαίως και θα πρέπει να προστατεύσουμε τους καταναλωτές ιδιαίτερα εσείς στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσετε μέχρι πού θέλετε να φτάσουμε για την προστασία, στο θέμα της προστασίας του καταναλωτή. Ναι, στην εναρμόνιση ώστε να τον περισσότεροι. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το θέμα της σχέσης μεταξύ φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόβλημα στο δίκτυο φυσικού αερίου μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και τα νάπαλιν. Επίσης η περιφερειακή διάσταση είναι κάτι το οποίο βρίσκεται απανταχού του κειμένου του κανονισμού. Έτσι θα πρέπει να εκφραστεί με συγκεκριμένου όρους η αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη δεν προκύπτει μόνο στις στιγμές, στιγμές κρίσης. Πρέπει να ενσωματωθεί στις πολιτικές των κρατών μελών αλληλεγγύη μεταξύ όλων των ε, φορέων και ενδιαφερομένων επιχειρήσεις, κρατημέλη, ρυθμιστές, TSO, οι πάντες. Και βεβαίως χρειάζεται και μια περιφερειακή διάσταση ενσωματωμένη σε αυτό το σύστημα και γι' αυτό εμείς σκαρφιστήκαμε το νη 1 Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί θα είναι η πιο χρήσιμη για να δούμε πώς και πού θα πρέπει να ενδυναμωθεί η περιφερειακή διάσταση, αλλά και βεβαίως θα αναλάβουμε το ρόλο μας ως διαμεσολαβητού μεταξύ των διαφόρων φορέων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Όπως είπε ο κ. Σπιώτη Πρόεδρε, πρέπει να Έχουμε ένα μοντέλο για την, ε, διάφορα μοντέλα για την ακρίβεια και να δούμε με προβολές στο μέλλον πώς αυτά τα μοντέλα θα ανταποκριθούν στις διάφορες κρίσεις. Ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να δώσω στην κυρία Κανιέτε το λόγο, η συγγήτρια από την ΕΜΚΟ. Πριν ε, τελειώνω, να δώσω το λόγο στον δικό μας εισηγητή. Κυρία Κανιέτε, ευχαριστώ για την υπομονή σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω την μητρική μου γλώσσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, εμπειρογνωμονές μας για την ε, πλούσια αυτή συζήτηση, γιατί πολλά από τα ζητήματα που συζητήσαμε στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς ακούστηκαν και εδώ πέρα. Δηλαδή θέλουμε ξεκάθαρο ορισμό του προστατευόμενου πελάτη. Πρέπει να είναι ρεαλιστικός, πρέπει να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, θα θέλαμε έναν σαφή ορισμό για τους ε, προστατευόμενους πελάτες ε, που να συμπεριλαμβάνει και τα νοικοκυριά και τα νοσοκομεία. Ε, γιατί αν πούμε πως όλοι οι πελάτες είναι προστατευόμενοι, τότε δεν είναι κανείς. Και εμείς ε, στην Επιτροπή μας λέμε πως πρέπει να αυξηθεί η ασφάλεια παραξιαρίου με τρεις τρόπους. Στις εταιρείες, στα κρατημέλη και στην κοινότητα. Οπότε πρέπει να ορίσουμε τον ρόλο και την ευθύνη των εταιριών σε καιρούς κρίσης. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τονίσουμε τον ρόλο των μηχανισμών της αγοράς και σε περίοδους κρίσης πρέπει να διασφαλίσουμε πως οι εταιρείες αυτές θα εργάζονται να δυνατόν περισσότερο και πως ε, μόνο ως ε, τελευταία λύση θα καταφύγουμε σε μέτρα εκτάκτου ανάγκης και τέλος κάτι για την ανταλλαγή πληροφοριών. Εμείς υποστηρίζουμε την Κομισιόν πράγματι πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαβούλευση με την Κομισιόν πριν ε, συναυθούν συμβάσεις με τρίτες χώρες ε, που επηρεάζουν την ε, προμήθεια αερίου. Τα μέλη της Επιτροπής μας θεωρούν πως αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στην οδηγία, όπως επίσης και η αλληλεγγύη και εννοούμε και την διασυνοριακή αλληλεγγύη και εντός της χώρας για να προστατευτούν οι πιο ευάλωτοι πελάτες και δεν πρέπει τέλος να ξεχνάμε πως ε, η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο δεν είναι μόνο τμήμα της ενέργειας πρέπει να έχουμε ένα κείμενο που θα αντικατοπτρίζει και τις ε, ανανεώσιμες πηγές καθώς ε, Επίσης ε, γιορτάζουμε και την 20η επέτειο από την πτώση του τείχους του Βερολίνου αλλά γιορτάζουμε ταυτόχρονα και την κύρωση της ε, συνθήκης ε, της Λισαβόνας αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα την απειλή ελήψεων φυσικού αερίου από την Ανατολή και πρέπει να προστατεύσουμε τους πελάτες μας να έχουμε μια σταθερή ροή αερίου και να γνωρίζουμε πως ε, ίσως το άμεσο μέλλον να αντιμετωπίσουμε κρίσεις. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αντιδράσει γρήγορα. Μας ενδιαφέρει λοιπόν ο κανονισμός αυτός ε, να εγκριθεί το στομότερο δυνατόν και είμαστε ικανοποιημένοι από την συνεργασία που είχαμε και για τη σημερινή συζήτηση επίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές που δέχθηκαν την πρόσκλησή μας και είναι πολύ καθυσχαστικό για μένα που διαπιστώνω ότι συμφωνώ με τις περισσότερες προστάσεις αυτών. Κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται και στο σχέδιο αναφοράς. Η πρώτη γραμμή άμυνας κατά τη διάρκεια της κρίσης είναι μια πλήρως ολοκληρωμένη και λειτουργούσα εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. Μόνο έτσι μπορέσαμε να υπερβούμε την προσφατή κρίση. Παρά τους περιορισμούς που υπάρχουν σε διαμφθοριακό επίπεδο. Εάν κατάλαβα καλά, κατά την περσινή κρίση το πρόβλημα δεν ήταν η έλλειψη φυσικού αέριου, αλλά οι φυσικοί περιορισμοί των υφιστάμενων διασυνδέσεων, αλλά και ο περιοριστικός χαρακτήρας πολιτικών συμφωνιών που ύψωσε εμπόδια στον δρόμο της ελεύθερης ροής του αερίου. Η Κομισιόν λοιπόν θέλησε να αντιμετωπίσει στη ρίζα τους τα προβλήματα αυτά. Και εμείς στο Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ούτε αυτούς που δεν δημιούργησαν προβλήματα αλλά που συνεισέφεραν στην εξέβεση λύσης. Εις ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών, οι φιλοξενούμενοι μας είπαν ότι η πολιτική θα πρέπει να βρουν τις λύσεις. Το μόνο μου σχόλιο είναι ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ πλήρως με την εκτίμηση του θέματος που αφορά την αντίστροφη των ροών και την σημασία της ε, περιφερειακής διάστασης αλλά και της ελαστικότητας για τα σχέδια αναδίπλωσης. Συμφωνώ με τη σημασία του θέματος της αποθήκευσης παρόλο που πιστεύω ότι αυτό το συγκεκριμένο θέμα, η αποθήκευση δηλαδή, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μιας αυτόνομης πρότασης λόγω της πολυπλοκότητάς του και για λόγους διαφανείας προστασίας του απορρίτου κτλ. Στο δεύτερο γύρο παρεμβάσεων σας ήσασταν πιο επίοικείς έναντι του κριτηρίου του νη 1. Το σημειώσαμε. Όμως, πολλοί ενδιαφερόμενοι από διάφορους χώρους προερχόμενοι θέτουν τεχνικά ζητήματα. Είναι πολύπλοκα και δεν θα τα συμπεριλάβω, πιστεύω ακόμα, στο πρώτο αυτό σκαρίφημα της ε, αναφοράς μου. Πάντως εγώ πιστεύω ότι το νη μείον 1 θα πρέπει να είναι ο βασικός παράγοντας επικουρικότητος για τα κράτη-μέλη, εφόσον κάθε εθνικό μοντέλο παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε ό,τι αφορά τη φύση, τα χαρακτηριστικά της αγοράς φυσικού αερίου, αλλά και ενεργείας γενικά. Για τον Ήμιον 1, προς το παρόν, το κείμενο θεωρώ ότι είναι πολύ ακαμπτό και δεν δίνει περιθώρια στην εφαρμογή της επικουρικότητας όπως θα έπρεπε. Ένα πολύ σημαντικό σημείο που έφεραν οι φιλοξενούμενοι μας σήμερα είναι ότι θα πρέπει να έχουμε ένα κοινό σύστημα το οποίο να είναι υποφελές για όλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το παγιώσουμε. Το πακέτο για την εσωτερική αγορά ενεργείας ήδη προβλέπει διαδικασίες μεταξύ των ρυθμιστών για διαμεθοριακή συνεργασία και υποδομές. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε συνεπείς με το περιεχόμενο του τρίτου πακέτου και αυτού του κανονισμού. Θα αποστείλω προς μετάφραση την Τετάρτη